I think we can start. Μπορούμε και να ξεκινήσουμε ίσως. Με έχω τη μεγάλη χαρά να υποδεχθώ τον Πατ Κόξ. Είναι πολύ γνωστός ως κοινοβουλευτικός, υπήρξε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για πολύ μεγάλο χρόνο βουλευτής και είναι τώρα συντονιστής για τον διάδρομο μεταξύ Σκανδιναβίας και Μεσογείου. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα για την παρουσία του Παρκόξ. Ξέρει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Για 10 λεπτά έχει το λόγο. for the opportunity to speak to you about the Ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας μιλήσω για αυτόν τον διάδρομο από τη Σκανδιναβία μέχρι την Μεσόγειο. Σας προτείνω στη σύντομη παρουσίασή μου να κάνουμε το εξή, Να σας μιλήσω για το σχέδιο εργασίας για αυτόν τον διάδρομο, να πούμε δύο λόγια επίσης για την διαδικασία που ακολουθείτε και θα σας μιλήσω για κάποια από τα αποτελέσματα και για ε, κάποια προγράμματα χρηματοδότησης που έχουν να κάνουν με αυτόν τον διάδρομο. Και επίση να σα πω δύο λόγια για τα επόμενα βήματα τα οποία προτείνουμε. Α, να, η διαφάνεια. Καθώς γνωρίζετε είχαμε την αφετηρία μας για αυτούς τους διαδρόμους. Και το 2014 όλοι οι συντονιστέ ορίστηκαν ή διορίστηκαν τέλο πάντων και αρχάσαν ένα άρχισαν να δουλεύουν και λάβαμε αυτή την επίσημη επιστολή του διορισμού μας και από τότε προχωρούμε σε κάποια συναντήσεις με τα κράτη-μέλη, με περιφέρειες επίσης, εταιρείε υποδομίες και άλλους εμπλεκομένους τόσο ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε τις επαφές και με εξωτερικούς συμβούλους για να προχωρήσουμε αυτά τα σχέδια των διαδρόμων και να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο είδους ε, συμφωνία στις βασικές μεταβλητές του τι θα τι διάδρομος. Θα σας πω πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλά είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις με ερετούς άρχοντες και με ευρωβουλευτές και με την Επιτροπή σας και με άλλους ευρωβουλευτές από τα λεγόμενα κράτη-μέλη, με μερική κυβέρνηση, ε, υπουργεία και τοπικές αρχές. Αυτός ο διάδρομος από Σκανδαλία μέχρι Μεσόγειο, εδώ περιγράφεται δύο λίγων. Σε αυτήν την διαφάνεια καλύπτει 7 κρατημένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, περνάει από τη Γερμανία, την Αυστρία, την ε, Ιταλία και μέσω Σικελίας καταλήγει στην Μάλτα. Επίσης νοτίως του Όσλο έχουμε την ε, σύνδεση του Όσλο με το Γκόντεμπουργκ. Και αυτό θα καλύψω. Οπότε είδατε ότι εδώ έχουμε καλύψει και 18 κόμβους και όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν από τον κανονισμό σας του 2013. Έχουμε επίσης 19 ε, αεροδρόμια πυρήνα και λιμένες πυρήνα 25. Επίσης θερματικούς ε, που συνδέουν δρόμους και Ρόδο ε, που αριθμούν 44 και επομένως είπαμε ότι μιλούμε για ένα διάδρομο που αντιπροσωπεύει το 27% του ΕΠ και το 16% της ε, ε, έκτασης. Τώρα, ο διάδρομος Ε, κατά ε, το πρώτο έτο λειτουργία θα έπρεπε να ε, υιοθετήσει κάποιε μεταβλητέ, κάποια κριτήρια με τον κανονισμό και να καλύψουμε λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρόμου κλπ. Και έτσι κάθε τρόπο μεταφορά θα έπρεπε να εξεταστεί αν συνάδει προ τον κανονισμό. Οπότε βλέπετε εδώ για τον σιδηρόδρομο ένα από τα κριτήρια είναι ο εξηλεκτρισμός του δικτύου, επίσης τα συστήματα ενέργειας, και πιο κάτω λέμε για το βάρος επί του άξονα. Το τέταρτο κριτήριο αφορά το μήκος των ε, ε που είναι 740 μέτρα και πέμπτο είναι το να ισχύει το σύστημα ERTMS αυτού του είδους το FES σύστημα παρακολούθησης των σιδηροδρόμων. Οπότε είπαμε ότι θέλουμε να καλύψουμε 9.000 χιλιόμετρα και όλα αυτά να δούμε αν συνάδουν προς τα κριτήρια. Και εάν έχετε ευνίες στο βράδυ να τσεκάρετε στο ίντερνετ τι γίνεται. Τι γίνεται και για αεροδρόμια, για ε, λιμάνια και όλα αυτά είναι εντελεχώς τα καθορίσαμε. Αν τώρα μια ματιά στο κατά πόσο αυτά συνάδουν με τα πρότυπα των διευρωπαϊκών δικτύων. Έχουμε εδώ πέρα κάποιες, ε, κάποιες προκλήσεις που έχουν επισημανθεί πρώτα πρώτα για, τον, ε, για, τους, δρόμους έχουμε ε, τις ε, συμφορήσεις και τα σχετικά μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με έργα υποδομής. Φερρυπίν, ε, τα πάρκιν και λοιπά. Όσον αφορά το τους λιμένες, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη έρευνα. Αλλά αυτό που κυρίως ενδιαφέρει από πλευράς της ξηράς, γιατί θα ασχοληθεί με τους αυτοκινητοδρόμους ο, ο Σίμψον είναι αυτού του είδους οι συνδέσεις με την ενδοχώρα. Επίσης για τα αεροδρόμια έχουμε τη συνδεσμένη μεταφορά ως προς τον ε, σιδηρόδρομο και όλα αυτά τα αεροδρόμια πυρήνα συνδεμένα με σιδηρόδρομο εκτός από τα 6 μικρότερα. Τέλος δε έχουμε αυτούς τους τερματικούς που συνδέονται, συνδέονται τερματικός τρένο με αυτοκινητόδρομο. Επίσης προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα για αυτόν τον διάδρομο και ποιοι είναι οι κρίκοι της σελίδας που έχουν πρόβλημα. Είπαμε ότι έχουμε το τούνελ ε, του, της διάβασης Μπρένερ. Και επίσης είδαμε ότι υπάρχει και η σταθερή σύνδεση του Φέρνερν και συνδέει το Αμβούργο με Κοπενχάγη προς Μάλμο και Στοχόλμη. Έτσι δε έχουμε τη γέννηση μιας καινούργιας μακροπεριφέρειας στην Ένωση. Ιδιαίτερα δε έχουμε προσέξει το πώς θα χρησιμοποιήσουμε το ERTMS. Θα σας τα πω σε λίγο. Όμως προς το παρόν είναι βαλωματική εφαρμογή του Άρα κάτι θα πρέπει να κάνουμε στην περίοδο αυτή που μας ενδιαφέρει, δηλαδή μέχρι το 2030. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα αναβαθμίσουμε. Έχουμε εδώ μια μακριά ε, λίστα, συνδέσεις ε, λιμένων, εναλλακτικά καύσιμα και ε, επίσης του σταθμού ανεφοδιασμού. Χρηματοδότηση, ισχύει το ένα σύστημα Αυτά πριν προχωρήσουμε σε κάποιο είδου εμπορική εκμετάλλευση που θα εξειδικευθεί στο μέλλον και θα αντιμετωπίσουμε επίση και τα σημεία συμφόρηση των κρατών μελών σε σχέση και με τα οδικά δίκτυα. Επίση, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε ποιε είναι οι ανάγκε για επενδύσει. Μέχρι τώρα για το SCANMED είπαμε ότι έχουμε 394 σχέδια και έργα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2030 για να πετύχουμε του στόχου μα. Είπαμε ότι οι συνολικές επενδύσεις για όλα αυτά, για τον διάδρομο, πάνε στα 144 δις ευρώ. Αυτό όμως καλύπτει μόνο το 73% που είπαμε πριν. Ε, οπότε αυτό δεν καλύπτει όλη την υπόθεση. Άρα το 144 δις το ποσό είναι ένα τμήμα των όσων χρειάζονται. 73% επομένως 100 αφορούν του δρόμους, 21% δρόμους, 3% λιμάνια και 3% ε, αεροδρόμια, ε, τερματικούς ε, τρένων και αστικούς κόμβους. Επίσης θα πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο προγραμματισμού εκτό από την επένδυση για το μέλλον. Τώρα να δούμε ποιε είναι οι βασικέ προτεραιότητε, όλα αυτά που είπατε εσεί στα πλαίσια των συζητήσεων για τον κανονισμό. Είπαμε λοιπόν, θα χρειάζονται κάποιε συνδέσει διασυνοριακέ. Αυτό είναι προσθέμενη αξία και είναι το θέμα κλειδί που ακολουθήσαμε του περασμένου 12 μήνε. Οπότε ξαναγυρίζουμε τώρα στην υπόθεση τη σύραγγας ε, του Μπρένερ και τη σύνδεση γιατί δεν ωφελούν οι συνδέσεις αυτές και τα τούνελ εάν δεν έχουμε καλή πρόσβαση. Οπότε γι' αυτό μας απασχολεί και συνεργαζόμαστε με τα μπλεκόμενα κράτη-μέλη. Τώρα όσον αφορά ε, τους λιμένες αυτές είπε ο Μπρέιν Σίμψον είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους. Και επομένω αυτό είναι η κοινή μας αρμοδιότητα το πώς θα υπάρξει επένδυση για το σύστημα ERTMS και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μακροπρόθεσμα υπόθεση. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα ε, όσον αφορά την πρόσληψη κάποιων συμβούλων σε αμέσως επόμενες εβδομάδες ε, γιατί θα πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση περισσότερα δεν χτίστηκε σε μια μέρα η Ρώμη. Οπότε πέραν τη οικοδόμηση κατασκευή χρειαζόμαστε να κοιτάξουμε και αυτό το θέμα. Επίση να δούμε τι γίνεται με το λογισμικό, το συνοδευτικό και επίση να δούμε τι μέτρα θα έχουμε για το θόρυβο, για τη βιωσιμότητα, για χρηματοδότηση οριζόντια ή εντάρσια, Θα χρησιμοποιηθεί και πόσο το τρένο και όλα αυτά θα συζητηθούν παράλληλα με την ανάπτυξη της υποδομής. Επίσης, στρατηγική επικοινωνία, πολύ σημαντικό, οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό και να σας πω και κάποια παραδείγματα. Τι κάνουμε όσον αφορά τον διάδρομο. Νομίζω ότι είναι εύστοχα αυτά τα παραδείγματα καλής πρακτικής στο ΔΕΜ πρόγραμμα εργασίας. Ε, συμφώνησαν τα κρατημέλη που καλέσαμε να μας ρίξουν κάποιες ε, ιδέες και να φτιάξουμε κάποια εργαστήρια με αυτές τις ε, ιδέες γιατί αλλιώς τον έχει κανείς Βρυξέλλες να τα συζητά και να γυρίζει πίσω και να ρωτιέται γιατί το έκανε δεν λέει τίποτα. Οπότε λέμε τώρα για κάποιους αξιόλογους οι οποίοι μιλούν σε άλλους αξιόλογους για να πετύχουν κάποια αξιόλογα πράγματα. Οπότε είδατε πώς μπορέσαμε να δώσουμε μια στο θέμα με αυτά τα εργαστήρια ιδέων. Πάρα πολύ καλή υποδοχή ε, ε, για αυτά. Είδαμε τι έγινε με, την, ε, με το σύστημα συγκοινωνία στη Σουηδία. Το Υπουργείο Μεταφορών μα δάνεισε κάποια ε, στελέχη και θα μα βοηθήσει. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο. Και επίση, ε, μακάρι να έρθουν και άλλοι εμπειρογνώμονε από τι κυβερνήσει. Εάν βέβαια θεωρούν τα κράτη-μέλη ότι έχει νόημα να κάνουν αυτή την κίνηση. Τώρα, όσον αφορά την διακυβέρνηση. Και όσον αφορά αποστολές. Κάνουμε τέσσερις τέτοιες ε, συναντήσεις. Έχουμε συγκροτήσει ομάδες εργασίας όπως για όλους τους διαδρόμους, για εσωτερικές πλωτές οδούς, για λιμάνια, για περιφερειακές αρχές. Και τα έχουμε πει με τον κύριο Φοντερ και με τον κύριο Χούμπερτς και είπαμε ότι κάναμε τέτοιες αποστολές και επισκέψεις τον αριθμό 21 από τον Μάρτιο του 14. Επίσης είχαμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, μια τέτοια μελέτη τέλος Δεκεμβρίου και όλα τα κρατημέλια ενέκριναν το πρόγραμμά μας. Και υπήρχε δε συνένεση ομόφωνη. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς και όλους όσοι θεωρούν ότι θα κάνουν παρόμοια πράγματα με παρόμοιο χρονοδιάγραμμα σε τέτοια ενδιαβάσεις Οπότε πρόεδρε και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα τώρα να σας τονίσω το πόσο, πόσο, πόσο βοηθήθηκα και εγώ και οι συνάδελφοι από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό ωφελεί και, τον κύριο, και τη συνεργασία του κύριου Χούμπερτ με τον κύριο Φάντερ Όλα αυτά για την προπαρασκευή ε, και την ε, εκτέλεση αυτών των αποστολών. Τώρα, όσον αφορά την χρηματοδότηση. Για να δούμε. 29 έκτου. Ο Επίτροπος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το Connecting Europe Facility. Και είναι το πιο μεγάλο πακέτο επενδύσεων που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο επενδύσεων από τότε που το 1994 ασχοληθήκαμε με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Με μεγάλη μου χαρά επίσης βλέπω ότι πάρα πολλά έργα και σχέδια υποστηρίχθηκαν για τον διάδρομο. Έχουμε 14 τέτοια έργα για το διάδρομό μας. Θα τα χρηματοδοτήσει η Κομισιόν και μιλάμε για 1,92 δις, δηλαδή 50% του συνόλου των εκταμιευμένων πόρων. Και δύο από τα μεγαλύτερα από αυτά είναι ε, αυτή η σύνδεση Δανίας Γερμανίας που είπαμε και το Μπρένερ μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας εκεί πήγε η του του λέοντος αυτής της χρηματοδότησης γιατί ακριβώ πρόκειται για το ότι θα λύσουμε θέματα διασυνοριακά ε, θέματα ε, συμφόρησης και είχαμε 146 πάλι εκατομμύρια τα οποία θα πάνε σε άλλα ε, έργα για δρόμους, για σιδηροδρόμους της πόλης, για ευθύς συνδέσεις και τέτοιε ιδέε. Επίση, έχουμε ένα σώρο σχεδίων τα οποία χρηματοδοτείται από οριζόντια προγράμματα. Αυτό για τι αρτηρίε τη θάλασσα και το ER, ERTMS. Και αυτό καλύπτεται από το σχέδιό μα. Και μιλάμε επίση τώρα για το σύνολο των 735 σχεδίων που υπέβαλαν. Ε, έτσι, έχουμε δώσει μόνο 276 όμως τελικά εγκρίθηκαν. Βλέπετε όμως πόσο τεράστιο είναι το ενδιαφέρον ούτω ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν έργα υποδομή για τι μεταφορές. Πάντως, Πρόεδρε, τέλος, θέλω να σας πω τι θα κάνουμε σαν τελευταία βήματα, επόμενα βήματα, το Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο πρόκειται να ε, προσλάβουμε αυτού του συμβούλου για να μας βοηθήσουν στην επόμενη φάση. Ε, έχουμε τις καλύτερε γραμμές από εσά και για το ΣΕΦ, ε, για τις προτάσεις σας, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Οι βασικοί εμπλεκόμενοι συμφωνούν, οπότε και θα συνεργαστούμε μαζί σας για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας και έτσι να δώσουμε κάποιες αυτές αποδείξεις για το πώς η Ευρώπη βελτιώνει το μέλλον μας, πετυχαίνει τους στόχους της μέσω της υποδομής των μεταφορών. Αν θέλετε μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Τώρα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις. Κυρία Βιρκούνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Πατ Κόξ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας να σας έχουμε εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Ο διάδρομος αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς διαδρόμους. Είναι ένας από τους μακρύτερους διαδρόμους στην Ευρώπη. Συνδέει το βόρειο και το νότιο τμήμα της Ευρώπης. Και για μένα που προέρχομαι από τη Φιλανδία βλέπω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο διάδρομος γιατί δίνει και μία δυνατότητα σύνδεσης προς, την, ε, προς τα σύνορα της Ρωσίας και πρόσβαση στη ρωσική αγορά. Δεν έχουμε τώρα και τόσο πολύ εμπόριο με τη Ρωσία και δικαιολογημένα. Αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι πολύ καλό να έχουμε σύνδεση και προς την ρωσική και ασιατική αγορά. Γι' αυτό ο σκανδιναβικό μεσογειακός διάδρομος είναι πολύ σημαντικός για την Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτός ο διάδρομος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πολυτροπικού διαδρόμου γιατί συνδυάζει αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας, ε, σιδηροδρόμους, αεροδρόμια και Είχα την ευκαιρία να ακούσω προηγουμένως μια παρουσίαση του Πατ Κόξ, αλλά αυτό πριν δημοσιευτεί ο κατάλογος των υποδομών του Connecting Europe Facilities. Θα ήθελα τώρα να δω εσείς πώς βλέπετε αυτόν τον κατάλογο. Ξέρουμε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πολλά από τα κονδύλια τα οποία αφορούσαν τα δίκτυα αυτά έχουν ε, ήδη δρομολογηθεί και από τη σκανδιναμική πλευρά υπάρχουν πολύ σημαντικά λιμάνια και σιδηρόδρομοι οι οποίοι θα πάρουν αυτά τα κονδύλια, επίσης ε, εγκαταστάσεις υγροποιημένου αέρα, αερίου και scrubbers, φίλτρων κτλ. Είναι σημαντικά, υπάρχουν τώρα δύο λείποντες κρίκοι που θα πρέπει αυτοί να χρηματοδοτηθούν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας ικανοποιεί η τωρινή κατανομή των, κομβ, των κονδυλίων αυτών και αν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα κύρια σημεία συμφόρησης με αυτή τη χρηματοδότηση. Ένα ακόμα ερώτημα. Είπατε το επόμενο βήμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι η κόμβη σε αστικές περιοχές. Για χώρες όμως όπως η Φιλανδία θα ήθελα να θέσω το ερώτημα το εξή. Ξέρουμε ότι φτάνουν μέχρι την νότια Φιλανδία. Η, η διάδρομη, η βόρεια Φιλανδία δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς τους διαδρόμους. Μπορείτε να φανταστείτε στο μέλλον να έχουμε συνέχιση των διαδρόμων και προς τα βόρεια γιατί είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε και ε, συνδέσεις με τον ακτικό κύκλο. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος. Ο Βιμ Φαντερ Κάμπ. Α, δεν ήθελες το λόγο. Τον ήθελες. Καλύτερα να ακούσεις τους άλλους συντονιστές πρώτα, λέει Εντάξει. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι από τη Βόρεια Σουηδία. Και με ενδιαφέρει φυσικά αυτός ο διάδρομος για τις προτεραιότητες για τις οποίες πρέπει να ληφθούν αποφάσεις τη 10η Ιουλίου. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τι προτεραιότητες που έχουν ήδη τεθεί για το, τη Βόρεια Σουηδία και τη Βόρεια Φινλανδία. Με αυτό δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όμω θα πρέπει να υπάρχουν links, σύνδεσμοι, όπω σωστά μα, είπε ο συνάδελφο. Ε, και θα ήθελα από περιέργεια να σα ρωτήσω και κάτι. Είστε συντονιστής. Πώς ακριβώς συνεργάζεσαι με τα κράτη-μέλη ούτως ώστε ε, να συντονίσετε τη συγχρηματοδότηση από πλευρά των κρατών μέλων. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω πώς μπορώ να επιτύχω, ε, παραδείγματος χάρη, με μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση για τη σύνδεση Όσλο-Κοπενχάγη, παραδείγματος χάρη, από πλευρά των Σουηδικών αρχών. Δεν είναι προτεραιότητα, αλλά για μένα είναι σημαντικό. Και μία άλλη ερώτηση. Πολύ ωραία αυτά τα εργαστήρια ιδεών. Μου φαίνεται ότι είναι εξαιρετική ιδέα, διότι όταν γίνονται πελούριες επενδύσεις στις υποδομές, ε, ε, εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι, πολλές γνώσεις ε, και συνέχεια χρειαζόμαστε νέες ιδέες. Τι πιστεύεις λοιπόν, πιστεύεις ότι μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω αυτή την πρωτοβουλία πέρα από αυτές τις περιφέρειες, πέρα από αυτούς τους διαδρόμους, δηλαδή αυτές οι ιδέες που γεννιούνται στα εργαστήρια μπορούν να μεταφερθούν, μπορούν οι πόλεις και οι περιφέρειες περιφέρειες ε, να αντιλήσουν αυτές τις ιδέες και έτσι να υπάρξει μεγαλύτερο δυναμικό καινοτομίας. Ευχαριστώ, η Γκίζινα Μάισνα. Ευχαριστώ. Εντάξει, μπορώ να λάβω το λόγο, ναι. Δεν ήμουν στην αρχή, γι' αυτό περίμενα να μιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι. Είχα ένα συγκεκριμένο ερώτημα για το διάδρομό σας κύριε Κόξ. Το, η σύραγγα λοιπόν στον Μπρένερ είναι πολύ σημαντική όταν όταν η σύνδεση ότι είναι πολύ σημαντική και θα ξεπεράσει και το Ωρεσούντ. Αλλά Ξέρουμε επίση εδώ και πολύ καιρό ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Δανία και Γερμανίας να υπάρξει μια σταθερή σύνδεση. Όταν γίνει λοιπόν αυτό, θα πρέπει να γίνουν και οι υπόλοιπε ενέργειε. Είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται. Αυτό μπορεί να είναι γερμανικές αρμοδιότητες. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει και αυτή η περαιτέρω σύνδεση. Μπορείτε να το επηρεάσετε αυτό. Και επίσης η διαδρομή Y η οποία θα συνδέσει το, τη Βρέμη, το Ανόβερο και το Χάμπουργκ. Έχουμε δώσει πολλά χρήματα στο, στη Γερμανία για το θέμα αυτό και τώρα υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Αλλά είναι αυτό που είπε ο συνάδελφο κ. Γιάννησεν. Ποιε είναι οι δυνατότητε να επηρεάσετε τι κυβερνήσει της Ελλάδος για να καταλάβουν ποια είναι η υποστέμενη αξία που μπορεί να προέλθει από αυτά τα σχέδια και χρειαζόσαστε την υποστήριξή μας. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Ένα περαιτέρω ερώτημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό <clears throat> να υπάρξει συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών σχέδιων. Πώς συνεργάζεστε με τον Brian Simpson, ο οποίος έχει να κάνει με τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας, ποια είναι η συνεργασία σας και επίσης σε ποιο βαθμό εσείς ως συντονιστής εμπλέκεστε στην στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες, χάρη Αδριατική, Ιόνιο ή Βαλτική. Αυτό θα είχε πολύ νόημα αν είσαστε συντονιστής να έχετε επαφή και με τους αρμόδιους για αυτές τις θαλάσσιες λεκάνες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Φαντερκάμπ. Πολύ ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Κόξ μας μίλησε ήδη για τα θέματα ε, επικοινωνιακής πολιτικής. Έχω θέσει το ίδιο ερώτημα και στους υπόλοιπους συντονιστές. Ε, ξέρουν τα πάντα οι Ευρωπαίοι πολίτες για τον Brexit, αλλά για τα δε χαμπάρι. Ξέρω ότι έχετε συνεργαστεί με δημάρχους, με συμβούλους, ε, με τους λαούς της Ευρώπης, αν μπορώ να το θέσω έτσι, έχετε μιλήσει, τους έχετε εξηγήσει. Δεύτερη ερώτηση. Τι γίνεται με την αδειοδότηση. Είναι αρκετά περίπλοκα αυτά τα προγράμματα και η βιωσιμότητά τους έχει υψηλές απαιτήσει, δηλαδή ε, απαιτήσει που τελικά αποφασίζονται και εγκρίνονται από, τις, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς ακριβώς, ποια, ποια πολιτική ακολουθείτε για την αδειοδότηση. Ε, και τρίτη ερώτηση είναι λίγο πιο τεχνική. Υπάρχουν διαφορές ως προς τη χρήση διαφόρων τμήματων του διαδρόμου. Παραδείγματο χάρη ανάμεσα στο Αμβούργο και στο Ανόβερο, φαντάζομαι στη Γερμανία είναι υψηλή συχνότητα οι επικοινωνίες. Υπάρχει διαφορετική ένταση, διαφορετική συχνότητα, ανάλογα με το ποιο τμήμα του διαδρόμου μας απασχολεί. Ε, για το ΕΦΣΙ τώρα, επειδή μιλούσαμε και για το ΣΕΦ και η συνάδελφός μου η Έλκα το ανέφερε, προφανώς η, το, το, η σύραγγα Μπρένερ και η σύνδεση ανάμεσα στη Γερμανία και τη Δανία σίγουρα θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη. Ε, μπορούμε στα πλαίσια του ΕΦΣΥ να ενεργοποιήσουμε την χρηματοδότηση. Τώρα έχουμε και ένα προσκεκλημένο από την ΕΚΟΝ. Παρακαλούμε, έχετε το λόγο. Κύριε Σάντ. Ε, θα ήθελα ε, να ρωτήσω τον ε, κύριο Κόξ, ε, επειδή είναι συντονιστής του προγράμματος, τι πιστεύει για την αποτελεσματικότητα των νέων υποδομών που προβλέπονται από τις κατευθύνες γραμμές των ΔΕΔ. Ε, αυτό το πρόγραμμα εργασίας ε, για το διάδρομο όπως και άλλα στην ίδια κατηγορία θα λειτουργήσουν ε, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί οικονομικής ανάπτυξης ανάμεσα στις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. οικονομική ε, σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προτεραιότητα για όλους μας ε, και ίσως ε, με αυτόν τον διάδρομο μπορούμε να έχουμε και καλύτερες εμπειρίες ώστε στην πράξη να επιτύχουμε σύγκληση ανάμεσα στις περιφέρειες. Θα ήθελα να ξέρω αν εσείς κύριε Κόξε ή άλλοι συντονιστές άλλων διαδρόμων έχετε σχέση με τις προτάσεις ε, του ΕΦΣΙ, ε, το Αμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, και του σχεδίου Juncker, γιατί ένας από τους δεδηλωμένους στόχους είναι η μεγαλύτερη σύγκληση. Κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ε, συναντήσατε συγκεκριμένες δυσκολίες ε, για τον συντονισμό των προγραμμάτων ανάμεσα σε περιφέρειες ε, που έχουν αποκλίνοντες αναπτυξιακού αναπτυξιακούς βαθμούς, για να το πω και πιο ξεκάθαρα, σε περιφέρειες του Βορρά και του Νότου. Ευχαριστώ. Παύλ Τελίτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πάντα αυτά που με είπε σήμερα και αυτά που ακούσαμε από άλλους συναδέλφους επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η νέα αντιμετώπιση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μπορεί να αποτελέσει μια επιτυχία. Και είναι η καλύτερη προσπάθεια που έχει γίνει για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις υποδομές μεταφορών στην Ευρώπη δεδομένων των περιορισμένων πόρων που έχουμε. ευχαριστώ και για την πλήρη σου έκθεση. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που τέθηκαν και έχει απαντήσει ήδη σε μερικά από αυτά που θα έθετα. Είναι πολύ καλό ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ εσού και του συναδέλφου σου από τους ε, αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας και όπως είπε και η Γεζίνα θα με ενδιαφέρε να ξέρω σε ποιο συγκεκριμένο επίπεδο από τη στιγμή που έχει εγκριθεί το ΕΦΣΙ, το σχέδιο Juncker, θα μπορούσατε να πείτε ότι επειδή χάνονται κάποια χρήματα από το Connecting Europe Facilities, θα ήθελα να ρωτήσω αν τα κάτι μελη έχουν δείξει ότι θα χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση αυτή να χρηματοδοτήσουν με το σχέδιο Juncker σχέδια τα οποία κανονικά θα ήταν στο Connecting Europe Facility. Στη δική σου περίπτωση του διαδρόμου πιστεύω ότι το Connecting Europe Facilities αντιμετωπίζει σχέδια διαφορετικού τρόπου από ότι το ΕΦΣΙ, το σχέδιο Juncker σε ό,τι αφορά την επιστροφή για τις επενδύσεις. Επίσης, ποια είναι η εμπειρία σου με τις μεταρρυθμίσεις θα ήταν αυτό ένα χρήσιμο εργαλείο ή απλώς ήταν υπερβολικά ψηλές οι προσδοκίες για το θέμα αυτό. Έχω δύο ερωτήσεις αλλά Έχουμε ήδη απαντηθεί από σένα. Ευχαριστώ. Ο Ντομινίκ Χρικέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω μία και μόνη ερώτηση. Υπάρχει ένα σημείο στον διάδρομο όπου διασταυρωνόμαστε με το δίκτυο της Βαλτικής που περνά από την Γερμανία και εκεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μελετά κάποια συμπληρωματικά οδικά έργα. Σημαντικά. Τι σκέφτεστε. Κάνουν συντονισμό κάποια ομάδα επαφής για το πώς θα γίνει αυτή η διασταύρωση των δύο τόσων στρατηγικών έργων εκεί. Κράμερ. Σε ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε τα θέματα τα διασυνοριακά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ακριβώ αυτά τα σημεία είναι αυτά τα οποία μα δίνουν την προσθεμένη αξία. Οπότε θα ήθελα τώρα να μου πείτε όσον αφορά τη, τα κρατημέλη τη εμπλεκόμενη χώρα, για πέστε μα, ε, εσεί ε, θα μπορούσατε να ασχοληθείτε πρώτα με τα σημεία τα διασυνοριακά. Ε, Ελφούρτη, Νιρεμβέργη, α πούμε, για τη Γερμανία. Πρώτα να κάνετε αυτά και μετά το υπόλοιπο υπάρχει κάτι το οποίο του παραχρόνου πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλά τι γίνεται με το Μπρένερ και σε σχέση με το Μόναχο εκεί. Δεν, δεν, δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται κάτι, δεν υπάρχει κάποια έγκριση. Μιλάμε όμω για ένα δι για τα εθνικά σχέδια. Αυτά έχουν εκταμιευθεί. Όμω τι γίνεται με τα σημεία τα διασυνοριακά που η Γερμανία δεν τα έχει καλύψει. Τι επομένω ε, ε, κίνητρα μπορείτε να δώσετε ε, κάποιο είδους ε, συμφωνία, δηλαδή να τους πείτε ότι θα πάρετε τα χρήματα μόνο εάν ασχοληθείτε και με την κάλυψη των διασυνοριακών περασμάτων, ας πούμε. Όσλο, Τρέλεμπορκ, Ροστόκ κλπ. Τώρα, Τρέλεμπορκ, Ροστόκ. Υπέροχη σύνδεση αυτή. Το Ροστόκ είναι ένα λιμάνι, αλλά και το Τρέλεμπορκ. Επομένω. γιατί κάνετε αυτή την παράκομψη, γιατί δεν κάνετε κάπως πιο ευθεία χάραξη, μια που είναι εντυπωσιακό αυτό. Γεζίνη μίλησε για αυτήν την ε, λευκή γραμμή. Αμβούργο, Βρέμι, Ανόβερο. Όλοι περνάνε από τη Σκανδιναβία μέσω Αμβούργου. Αυτό μας οδηγεί εκεί σε εμπλοκή, σε, σε, σε συμφόρηση. Άρα βρέστε κάτι. Τραβημούντε, Τρέλεμπορντ, το Φέρνμπελτ και εκεί θα πρέπει κάτι να γίνει. Για το Φέρνμπελτ έδωσε την έγκριση η Γερμανία. Είπε ότι αν θέλει να δώσει την άδεια να πληρώσει η δανειζική κυβέρνηση, εμεί πάμε πάνω. Αλλά η Γκεζίνε είχε δίκιο σε αυτό που είπε. Τι είπε ο είπε ότι είναι υπέρ του έργου εκεί. Μιλάμε για μία γραμμή σιδηροδρομική και δύο αυτοκινητοδρόμους. Ε, γιατί όπως μάθαμε στο σχολείο η αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο πιο αδυνάτος κρίκος της. Και έχουμε και το Connecting Europe Facility η Δανία. Από το Göteborg στο Νίκοπινγκ για να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε τη γραμμή που είναι 40 χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είχαμε τελικά μονάχα ένα τρίτο των χρημάτων που είχε προτείνει αρχικά η Δανία. Η Δανία είχε δημιουργήσει μια μεγάλη συζήτηση, αλλά ήταν και το θέμα τι θα κάνανε οι άλλες χώρες. Μήπως ε, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη χρηματοδότηση από τα κρατη Τι γίνεται αν Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν τις αντιδρήσεις από τα κρατημέλη, γιατί το πιο πρώτο ήταν να υπάρχει μια σύνδεση από το Τρέλεμπορκ στο Ρόστοκ. Και κάτι ακόμα, ναι είχα να πω κάτι και για τις διαμεθοριακές συνδέσεις. Πριν από 15 χρόνια έγινε ένας αυτοκινητόδρομος που περνούσε τα Πυρηναία και έφτανε στα γαλλικά σύνορα και εκεί υπήρχαν μονάχα επαρχιακές οδοί. Και τέτοιο πράγμα, είπε η Κομισιόν, δεν θα ξανακάνουμε. Από τη μια μεριά να υπάρχει ένα αυτοκινητόδρομο, ο οποίο είναι χρηματοδοτημένο κατά 50%, αλλά χωρί καμία σύνδεση από την άλλη πλευρά. Το φήμα Μπελτ λοιπόν θα μπορούσε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα, εάν δεν υπάρχει αυτό το τούνελ το οποίο συνδυάζεται με αυτό το φήμα Μπελτ. Και θα ήταν πολλά τα χαμένα λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη του Κοινοβουλίου για την ευρεία ποικιλία απόψεων που διατύπωσαν. Ευχαριστώ αυτού που έχουν δώσει και την υποστήριξή του σε αυτό το εγχείρημα και θα σα ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτό σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, αν είμαι ικανοποιημένο. Σε ό,τι αφορά την, ε, τα κονδύλια που μου δόθηκαν. Ήταν 730 ε, σχέδια για 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά Ήδη κάποια 200 πόσα από αυτά είχαν ε, θεωρηθεί ότι είχαν επιλεγεί και μόνο 276 περαιτέρω ενεκρίθησαν. Ένα το οποίο ήταν από τα πρώτα σχέδια ήταν ήταν ένα τούνελ το οποίο ε, επελέγει όπως το τούνελ του Μπρένερο. Για το Φέμενβέλτ ήταν έκτος των κατάλογο των 276 σχεδίων για να είσαι έκτος είναι ήδη θετικό και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στη συζήτηση ακόμα και αν υπήρξαν κάποια σχετικά σχόλια. Για το Μπέλτ 589 εκατομμύρια ευρώ πήρε αυτό το γύρο κατανομής κονδυλίων. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η σύνδεση Φέρμαν Μπέλτ θα παραταθεί και πέραν αυτής της σειράς κονδυλίων. Γιατί τα κονδύλια αυτά φτάνουν μέχρι το 2019 δεν υπάρχει κανένα σχέδιο το οποίο να έχει χρηματοδοτηθεί για το 2020. Αν αρχίσει λοιπόν να λειτουργεί, τότε η σταθερή σύνδεση Fairman Λίξ μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο, να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή, ώστε μέχρι να δούμε τις περαιτέρω προσκλήσεις στον επόμενο γύρο και όταν έχουμε το νέο Connecting Europe Facilities, όταν έχετε ένα νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, θα μπορέσει να συνεχιστεί. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ε, εκκίνηση και πιστεύω ότι αυτό το οποίο το, ξεκι... το ξεχωρίζει από το Μπρένερ είναι ότι το Μπρένερ είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα λοιπόν τα οποία υπάρχει λοιπόν μεγάλη ευκαιρία να είσαστε ικανοποιημένοι που ήρθε έκτο από τα 276 και ας κατανοήσουμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Αναφέρθηκε λοιπόν το θέμα της σύνδεσης με τη Ρωσία. Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι ήταν σημαντικό σημείο έμφασης με τις αρχές της Φιλανδίας και αν αφήσουμε τα γεωπολιτικά προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει, υπάρχει μεγάλη προσήλωση στα θέματα τα περιβαλλοντικά στη Φιλανδία για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συνδύσεις και το να υπάρχουν αυτές τις συνδέσεις στα σύνορα της Ρωσίας και να μπορεί κανείς να προχωρά προς τα νότια. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τον διάδρομο Σκανδιναβίας με την ε, ε Μεσόγειο. Για να έρθω στο θέμα που αναφέρατε για την Βόρεια Σουηδία και Βόρεια Φιλανδία. Ο διάδρομος σταματάει στο νότιο τμήμα των χωρών αυτών, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την οικονομική του βιωσιμότητα. Προφανώς θα γνωρίζουμε αυτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι άλλες περιοχές περιλαμβάνονται στο συνολικό πλαίσιο, στο συνολικό δίκτυο και ούτως ή άλλως εμείς δεν θεωρήσαμε ότι έχουν αποκλειστεί από αυτά και ότι δεν μπορώ σαν συντονιστή να συναντήσω του εμπειρογνώμονε για να μελετήσουμε και τα θέματα αυτά. Κάποιε από τι μελέτε οι οποίε γίνονται λοιπόν έχουν σαν στόχο να συνδέσουν τι περιοχέ παραγωγή του Αχρικού με τα νότια λιμάνια τη Σουηδία και τη Φιλανδία και του καημού του. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι δεν περιλαμβανόμαστε στο σχέδιο αυτέ οι περιοχέ, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έχουμε λεπτομέρειε οι οποίε θα οριστικοποιηθούν και έχω σχέδια να πάω στη Βόρεια Σουηδία προσκλήσει μια ομάδα δήμων που έχουν ήδη κάνει μεγάλες προσπάθειες για να κάνουν σαφείς τις ανάγκες τους παρά το γεγονός ότι δεν είναι μεγάλη η επιβατική κίνηση η κίνηση του φορτίου χίδη είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήταν πάρα πολύ σύντομο να, σημαντικό να έχουμε αυτήν την σύνδεση για τις πόλεις όπως είπατε έχουμε ένα μεγάλο πανόραμα 9.000 ε, χιλιόμετρα τρένου και 4.000 αυτοκινητοδρόμων θα ήταν παράλογο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Το θέμα λοιπόν του να έχουμε μια σωστή ε, συγκέντρωση των προσπαθειών είναι απαραίτητο. Γι' αυτό εγώ έχω πλησιάσει και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για να μας φέρει σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Δεν είμαστε ίσως αυτοί που έχουμε τους περισσότερους πόρους, αλλά είναι χρήσιμο να έχουμε μια επαφή μαζί τους. Κάναμε κάτι τέτοιο στο Μάλμε και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν και τους άλλους να συμμεριστούν την ευθύνη για τα θέματα αυτά. Για το Fairman Belt και απαντώ τα ερωτήματα για, ε, ε, για τις, ε, την επιρροή στον γενικό κόλπο εκεί πέρα της περιοχής, επειδή τέθη το θέμα αυτό, θα χρησιμοποιήσω το Φέρμαν σαν ένα παράδειγμα. Από τη δική μας άποψη, για να το κάνω σαφές, αν έχουμε μια σταθερή σύνδεση, δεν είναι ακριβώς η καλύτερη λύση. Ως Ιρλανδός είπα, είπα ότι είναι σαν να έχουμε ένα pub χωρίς μπύρα. Για τους Ιρλανδούς αυτό δεν είναι πολύ θετικό. Και τουλάχιστον με ακούσανε, γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό το επιχείρημα. Κάνουμε συνεχείς προσπάθειες, προσπαθούμε να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ αυτής της σύνδεσης σε κάθε επίπεδο. Όταν έχουμε σε επαφή με τον κύριο Ντόμπριντ, με τους υπουργού ε, των κρατηδίων στα, στη Γερμανία, όταν συναντώ το DB το Deutsche Bank, αυτό είναι επιτάπητος. Όταν μιλάω με τους συντονιστές που εμπλέκουν και αρμοδίους της κοινωνίας των πολιτών, πάντα μιλάμε για αυτήν τη σύνδεση. Τον Οκτώβριο θα πάμε στο Schleswig Holstein και θα μιλήσουμε με όλους τους αρμόδιους για να τονίσουμε τη σημασία αυτής της σύνδεσης. Και σε ό,τι αφορά το λεπτομεριακό έθος, η εταιρεία Fairmark Belt AS στην Δανία, η αρμόδια ε, επιχείρηση, κάνει πολλές προσπάθειες για να μπορέσει να πάρει τις απαραίτητες άδειε, Η διαδότηση βέβαια είναι πολύπλοκη και χρειάζεται χρόνο, αλλά έχουν προετοιμαστεί πάρα πολλά πράγματα για να αντιμετωπιστεί και το γερμανικό τμήμα αυτή τη σύνδεση και να δοθούν οι απαραίτητε άδειε. Η Φέρμαν ΕΕΣ e έχει δώσει απάντηση σε διάφορε ερωτήσει που τέθηκαν με 11.000 σελίδε κειμένου και ανάλυση. Έχουμε πάρει επίση και συγχρηματοδότηση. Έχουμε δώσει συγχρηματοδότηση για μελέτε. Επομένω εμπλεκόμαστε. Δεν συνδέω βέβαια τι μελέτε με το τελικό, τελική προσφορά για τι υποδομέ, αλλά θέλουμε να, έχουμε, να πιάσουμε τόπο τα χρήματά μα. Και το τελευταίο που θέλω να πω για τη Γερμανία και το θέμα παραγωγικά του Μπρένερο κτλ. Γιατί πολλοί διάδρομοι περνάνε από τη Γερμανία. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα είναι το νέο σχέδιο της ε, ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τις μεταφορές που θα δώσει προτεραιότητα μέσα στη Γερμανία για τα θέματα αυτά. Ιδίω εσείς που είσαστε Γερμανοί ξέρετε ότι υπήρξε μια τεράστια συζήτηση μέσα στη Γερμανία για τα θέματα αυτά αφήνοντας την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση προς το παρόν από τη Ομοσπονδία Βιομηχανιών κτλ. Είπανε ότι υπάρχει πραγματικά υποχρηματοδότηση που έχει να κάνει με την διατήρηση των υποδομών και την ανάπτυξη νέων υποδομών. Βλέπω λοιπόν, και αυτή δεν είναι δική μου ανάλυση, είναι κάποιο άλλο. Όλα αυτά είναι τμήματα μιας ευρείας συζήτησης. Χρειαζόμαστε πράγματι την ε, υποστήριξή σας. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα της κυρίας χτυπήστε πόρτες, μιλήστε με τον κόσμο. Δεν έχει νόημα να πούνε όλοι ότι θα συνεργάζονται μαζί μας, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Η συνεργασία με τον Brian Simpson. Ναι, κάθε φορά που επισκεφτόμαστε ένα λιμάνι και έχουμε επαφή με αυτούς, ενημερώνει τον Simpson και υπάρχει αυτή η συνεργασία για την λιμενική στρατηγική θα ακούσουμε και τις απόψεις των Υπουργών Μεταφορών της Σκανδιναβίας για να έχουμε μια συγκεκριμένη συνεργασία για τις επικοινωνίες σε γέννη, πέραν αυτών που είπα για το τούνελ του Μπρένερο λοιπά. Ένας από τους εμπειρογνώμονες που θα βοηθήσει την Κομισιόν θα είναι αρμόδιος σύμβουλος για τα θέματα επικοινωνίας. Θα ήταν χρήσιμο να ακούσετε και για αυτό το θέμα, αλλά σε πιο γενική βάση να σας πω ότι πιστεύω ότι δυστυχώς το CF και το TNT είναι άγνωστα στον ξένο, στο, στην κοινή γνώμη, δυστυχώς. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοούν τη σημασία των σχεδίων αυτών σε σχέση με το τι μπορούν να επιτύχουν. Ο μόνος τρόπος που γίνεται γνωστό αυτό το μήνυμα είναι με το να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη στην Ευρώπη για να μπορέσει να προωθήσει αυτές τις πολιτικές. Η, ο δρόμος, η διαδρομή Y, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ίσως υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση, αλλά η σύνδεση Βρένερο, <clears throat> Ανόβερο, Αμβούργο, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι είναι υπερβολικά υπερφορτωμένη. Για την συγχρηματοδότηση δεν έχω ένα σύνολο από σχέδια τα οποία θα αφορούν. <coughs> Χρειαζόμαστε να έχουμε φυσικά κάποια έσοδα τα οποία θα ε, αποσβέσουν το κόστος των σχεδίων. Αυτό θα ισχύει ίσως για τα συνδεδομικά δίκτυα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας κατάλογος σχεδίων που προσπαθεί να δει τι μπορεί να λειτουργήσει και για τη Μάλτα. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Να σας πω για τα θέματα σύγκλησης Βορρά και Νότου. Ναι, υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, υπάρχουν θέματα μεθοδολογίας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και έχω να αντιμετωπίσω άλλες κυβερνήσεις που έχουν πολλά προβλήματα, όχι επειδή δεν θέλουν να προχωρήσουμε, όχι επειδή δεν θέλουν να έχουν συνδέσεις, αλλά επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν από τα κριτήρια του Μάστριτ για να κάνουν τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις. Όλα αυτά λοιπόν να ξεπερνάνε. Θα ήθελα να υπάρξει η, η χρηματοδότηση ώστε και αυτό μπορεί να γίνει αν γίνει δεκτή η ιδέα ότι η χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων δεν θα πρέπει να μετρά στους κανόνε του ελλείμματο. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο πρόβλημα. Τα άλλα ερωτήματα τώρα. Ο Πάβελ <clears throat> αναφέρθηκε στα θέματα της, των εσόδων. Είναι απαραίτητο να έχουμε σωστή επικοινωνία και να έχουμε σωστή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων και να δημιουργήσουμε και μια μεγαλύτερη συνένεση για τα θέματα αυτά. Όλοι έχουν το ίδιο σχέδιο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά σε σχέση με το σχέδιο το οποίο πήγε στο Βερολίνο, στην Κοπεχάγη, στη Ρώμη ή στην Βαλέτ. Επειδή όλοι έχουν πει ναι, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια συνένεση, έμεση συνένεση. Και το ερώτημα του Ντομινίκ Κρικέ για τα σημεία τομή των ε, δικτύων και το πώς μπορούν να συνδυάσουν διάφορα σχέδια, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πέρσι οι συντονιστές βρεθήκανε 6-7 φορές και ίσως περισσότερες από 6-7. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας και πρόεδρε για τα διαμεθοριακά στοιχεία μεταξύ του Μονάρχου και του Μπρένερ. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι περιμένουμε το σχέδιο μεταφορών από την ε, γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήρθαμε με την εκτελεστική επιτροπή της Deutsche Bahn στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και είπανε ότι εξαρτώνται από την ύπαρξη δημοσίων χρηματοδοτήσεων. Αυτή τη στιγμή το μοντέλο που ακολουθείται δεν περιλαμβάνει ιδιωτικό χρήμα ή συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού. Αυτό μας ξαναγυρίζει στο γερμανικό σχέδιο μεταφορών. Είναι κυκλικό λιγάκι το επιχείρημα, αλλά εμεί περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες. Τέλος, σε σχέση με τις αμοιβέ προσδοκίες, αν μπορώ να το θέσω έτσι, επειδή όλοι έχουν το ίδιο σχέδιο, επειδή όλοι είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν αυτή τη συνένεση, επειδή όλα τα κράτη-μέλη με την εμπειρογνωμοσύνη τους για πρώτη φορά για πρώτη φορά από το 1994 συμφώνησαν τη χρηματοδότηση που ζήτησε η Κομισιόν με καμία αποχή, κανένα opt-out, κανένα να πει κάτι αντίθετο, είναι πραγματικά μια πρωτιά. Και αυτό δείχνει ότι με ένα σωστό μοντέλο, σωστό κανονισμό, σωστή χρηματοδότηση, μπορούμε να έχουμε μια αυξανόμενη συνένεση για πρώτη φορά στην ιστορία των Τέντι, των διευρωπαϊκών δικτύων, κανένα κράτος μέλος δεν στράφει εναντίον κάποιας από τις 276 προτάσεις. Αυτό είναι μεγάλη πρωτοτυπία, δείχνει ότι υπάρχει μια νέα κοινή ευφυΐα για το πώς θα φτιάξουμε το κοινό μας μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόξ. Πατ και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον. Προτού συνεχίσουμε τώρα, να σας υπενθυμίσω ότι ο Γιώργ Λάιφριτ έχει φύγει από την Επιτροπή Μεταφορών γιατί έχει γίνει υπουργό στην ε, χώρα του και η Καρολίν Γκράσμαν Χάιν είναι τώρα α, αντικαταστάτριά του και είναι αναπληρωματικό μέλος. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Να, Παρός πάνω. Ich begrüße jetzt σε χαιρετίζουμε λοιπόν. Καλώ ήλθε. Ήταν υπουργό μεταφορών στη Γερμανία και τώρα είναι ο πρόεδρο τη Επιτροπή η οποία εξασφαλίζει ότι θα μπορέσει να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή και είναι συντονιστής για το διάδρομο Βαλτικής Αδριατικής. Κάτι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που είναι εδώ παρόν είναι ο συντονιστής, όπως είπα, για το διάδρομο Βαλτικής Αδριατικής. Το σχέδιο δράσης το ξέρετε, έχει ήδη διανεμηθεί. Κύριε Μπότεβιξ, σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας, την ευγενική παρουσίασή σας. κύριε και κύριοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να εμφανιστώ ενώπιόν σα ω συντονιστή του διαδρόμου Αδριατική Βαλτική και να σα παρουσιάσω το σχέδιο δράσης μα. Και επίσης να κάνω σαφές ότι αυτός ο διάδρομος έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τη σύνδεση των διαφόρων δικτύων μεταφοράς στην Ευρώπη. Χαίρομαι που μονάχα <clears throat> μετά από ένα χρόνο, δηλαδή πριν από ένα χρόνο μου δόθηκε η εμπιστοσύνη της Επιτροπής σας για να αναλάβω το ρόλο του συντονιστή αυτού. Έχω τότε κάπως ασαφείς ιδέες, αλλά τώρα μπορώ να σας πω ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουν συγκεκριμενοποιηθεί πολύ περισσότερο όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω τα κύρια στοιχεία του σχεδίου δράσης μου, που έχουν κριθεί θετικά από όλα τα κράτη-μέλη και έχουν πάρει μια θετική υποστήριξη. Και αυτό υπενθυμίζει λιγάκι κάτι που είπε και ο Πατκόξ στη δική του παρέμβαση, ότι η συνεργασία στην Ευρώπη επί τη βάση της εμπιστοσύνης είναι η βάση της πρόοδου. Επιτρέψτε μου όμως να σας παρουσιάσω τον διάδρομό μου, ο Βαλτικός Αδριατικός Διάδρομος, όπως μπορείτε να δείτε στο γράφημα, στο χάρτη, συνδέει την Βαλτική με την Αδριατική και περνάει από έξι Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Σλοβενία, Ιταλία. Ο διάδρομος αυτός ξεκινάει από τέσσερα λιμάνια στην, ε, στο Σετσίν Σινούς, Γδίνια και Ντάνσκ μέχρι το αδριατικό λιμάνι της Ραβένας, της Βενετίας, της Τεριέστης και του Κόπερ. Πάνω από 4.200 χιλιόμετρα σιδηρόδρομο και 3.500 χιλιόμετρα οδικών αξώνων συνδέονται, αυτού, τι αυτές τις περιοχές, 13 αεροδρόμια, 13 αστικοί κόμβοι, 10 λιμάνια, και αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί έχουμε όλο και μεγαλύτερη εμπορευματική μεταφορά στην περιοχή είναι οι 30 ε, πλατφόρμες επιμελητίας κατά την, στο μήκος αυτού του διαδρόμου. Όλα αυτά συνδέονται με τις προδιαγραφές του, των διευρωπαϊκών δικτύων. Υπάρχει βέβαια μεγάλη πρόκληση στα τμήματα που είναι μεθοριακές περιοχές. Θέλουμε να ευνοήσουμε την, ε, τη συνδρομική μεταφορά στον τομέα της Βαλτικής και της Πολωνίας και στις άλλες περιοχές να ενισχύσουμε τις μεταφορές με δρόμους. Καταρχήν, είναι πολιτική προτεραιότητα η μεταφορά με σιδηρόδρομο. Το άρθρο 12 του κανονισμού των TNT θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ε, μεταφορά με σιδοδρόμους, τα λεγόμενα 10T standards. Εδώ υπάρχει μια σειρά από προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μαζί με τα εμπλεκόμενα αλλά και μαζί με όλους τους εμπλεκομένους. Εκτός λοιπόν από τα τμήματα τα οποία περνάνε τα σύνορα μεταξύ Μπαρτισλάβας και Βιέννης, είναι συνδέσεις οι οποίες θα έχουν και επιβατικό χαρακτήρα, θα πρέπει να ηλεκτροδοτηθούν τελείως, να γίνουν ηλεκτρικές γραμμές. Αλλά έχουμε τρία διαφορετικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύω και πρέπει να εξασφαλίσουμε την διαλειτουργικότητα τα οποία εμποδίσουν τις πολυσυστημικές ατμομηχανές, μάλλον μηχανές κίνησης να λειτουργούν. Επίσης υπάρχει το ελάχιστο φορτίο ανάξονα 22,5 τόνων. Μόνο 10% των υποδομών μπορούν να εξασφαλίσουν αυτήν την ε, προδιαγραφή και ιδίως στην Πολωνία και στην Σλοβενία. Για την ταχύτητα για τα εμπορικά τρένα υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες ε, διαφορές. Στην Πολωνία και στη Σλοβενία ιδίως υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της υποδομής περίπου 30% που δεν είναι συμβατό με την προβλεπόμενη ταχύτητα των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Για το μήκος των τρένων, και εδώ είναι τα πράγματα πιο δύσκολα, για το μεγαλύτερο μέρος του διαδρόμου 84% δεν φτάνει το <clears throat> μήκος το οποίο προβλέπεται 740 μέτρα και αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Για το σύστημα ERTMS δεν χρησιμοποιείται ακόμα σε αυτή, την, σε αυτή την περιοχή εκτός από ένα τμήμα στην Αυστρία. Δεν έχει τεθεί λοιπόν γενικά σε λειτουργία και επομένως είμαι σε επαφή με τον συναδελφό μου ο οποίος είναι αρμόδιος για την οριζόντια εφαρμογή του ERMTS γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητο εδώ πέρα να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα σηματοδότησης και ασφάλειας. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν ένα σημεία συμφόρηση που πρέπει να ξεπεραστούν και έρχομαι στο επόμενο ε, σημαντικό σημείο. Τα περισσότερα από τα προβλήματα αφορούν έξι ε, και δύο οδικές διαμεθοριακές διέλευσεις. Εδώ πρέπει να υπάρξει σημαντική βελτίωση για τη βελτίωση της συνδρομικής υποδομής. Είναι στα πολωνικά σύνορα από την Οπόλα στην Όστραβα και από το Κατόβιτσε προς την Όστροβα. Επίσης στα σύνορα Αυστρία και Σλοβακίας μεταξύ Βιέννη και Μπρατισλάβας έχουμε το τρίτο σημείο συμφόρησης πολυνοσλοβακικά σύνορα μεταξύ Κατόβιτσα και Τσίλινα, επίσης μεταξύ του Γκράτς και της Αυστρίας μεταξύ, και, του Μάριμπορ και επίσης Λουμπλιάνα Τεργέστη και ένα κόμμα στη Σλοβενία. Όλα αυτά φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικά. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε την απαραίτητη πρόοδο για τα θέματα αυτά. <clears throat> Αλλά ας έρθω και πάλι στα θέματα των οδικών ε, αξώνων εξακολουθούν να υπάρχουν δύο τμήματα συνοριακών διελεύσεων Κατόβιτσε και Στσίλινα στη Σλοβακία και επίσης το Μπρον με την ε, Βιέννη. <clears throat> Κυρίες και κύριοι, έχουμε και περαιτέρω προκλήσεις. Υπάρχουν δύο λεγόμενοι ελίποντες ε, κρίκοι σε αλπικές διελεύσεις πρωτογεννατούλες τους Αυστριακούς, στις Αυστριακές Άλπες, το Γκράφινσταν στο Βέλμισετς και το τούνελ από τον Κλόντιν στη Ζούτσουσνα. Όλα αυτά λοιπόν τα τούνελ θα μπορούσαν να κάνουν πιο σύντομες τις, τις και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των μεταφορών. Αλλά υπάρχουν και πολλά ε, θέματα που έχουν να κάνουν μεταξύ Πολωνίας και Σλοβενίας. Στην Πολωνία και στη Σλοβενία μάλλον πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις και στην Σλοβακία για τη διέλευση της Πολωνίας-Σλοβακίας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά τα οποία πρέπει να κάνουμε κυρίες και κύριοι. Πιστεύω όμως ότι έχει κάθε νόημα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο αυτούς τους διαδρόμους. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για το μέλλον γιατί όχι μονάχα έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα πηγαίνουν θετικά, αλλά και η εμπειρία μου από την εργασία μου δείχνουν ότι όλα τα κάτι μελη κάνουν μια προσπάθεια να υπάρξει ένα γενικά συμπεφωνημένο σχέδιο δράσης, το οποίο θα ακολουθηθεί και στο μέλλον. Από τα σχέδια αυτά, τα 350 σχέδια τα οποία έχουν εντοπιστεί για την ανάπτυξη του διαδρόμου μέχρι το 2030, ε, είναι αποφασιστικό χαρακτήρα αυτά τα σχέδια, εκπροσωπούν επενδύσεις 60 περίπου δισεκατομμύριων ευρώ. Και πάλι η προτεραιότητα είναι η σιδηροδρόμη, περίπου τα 50% πηγαίνουν για την σιδηροδρομική υποδομή και εκεί βρίσκονται και μεγάλες προκλήσεις, 30% για οδικές υποδομές. Εδώ απλώς για να κλείσουμε ορισμένα σημεία που αποτελούν και για το πέρασμα των συνόρων, 12% για τους λιμένες και 6% για τα αεροδρόμια, για τους τερματικούς αθμούς ε, ε και τους αστικούς κόμβους. Έχουμε λοιπόν μεγάλες προκλήσεις χρηματοδότησης και ελπίζω ότι για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο θα υπάρξει και πάλι μια, ένας τριπλασιασμός των, επενδύσεων στον τομέα αυτό, αλλά ακόμα δεν έχουμε αρκετά χρήματα, πρέπει να κάνουμε μια ιεράρχηση προτεραιότητα. Θα πρέπει να υπάρξει σταθερότητα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο αυτές τις υποδομές. Όσοι συντονιστής λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήθελα να υποστηρίξω τα κράτη-μέλη και τις περιοχές όπου υπάρχουν οι υποδομές για τα θέματα αυτά. Το σχέδιό μου λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα μαζί με τα κράτη-μέλη έχουμε θεσπίσει πέντε προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα είναι οι υποδομές σε διαμεθοριακές συνδέσεις και για οδικές και συνδροδομικές συνδέσεις. Εδώ είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε δυνατή μια ευρωπαϊκή δομή δικτύων. Ως Ευρωπαίος συντονιστής θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε ενδελεχώς με τα κράτη-μέλη για αυτές τις συνδέσεις για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον καλύτερο συγχρονισμό των ενεργειών και θέλουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στο σχεδιασμό των σχεδίων από τις δύο πλευρές ώστε να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ τους. Είναι φανερό ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κοινή δράση. Δεύτερον, θέλω να τονίσω και πάλι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε και να προωθήσουμε τις διελεύσεις των Άλπαιων στην ε, Αυστρία. Υπάρχει ακριβώς το θέμα αυτών των ε, σχεδίων για σύραγγες στην ε, Αυστρία που έχουν μεγάλη σημασία, αλλά πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Και με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει μεγάλη, μεγάλο κέρδος χρόνου, αλλά θα γίνουν και πιο ελκυστικές αυτές οι διαδρομές για τις εμπορευματικές μεταφορές. Τρίτον, η σύνδεση μεταξύ λιμένων και ενδοχώρας, το τελευταίο μίλι όπως λέμε, εδώ θα πρέπει να σας υπενθυμίσω, μίλησα με την κυρία Μπούλς και της το παρομοίωσα αυτό με, τους, με τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Είναι πάρα πολλά τσίπα τα λιμάνια τα οποία δεν έχουν καμία σύνδεση με λιμένες και έχουν μονάχα μία σύνδεση με αυτοκινητοδρόμους. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό θα αλλάξει. Τέταρτον, θα πρέπει να δώσουμε σημασία στους, ε, στους ε, αστικούς κόμβους που είναι πολύ σημαντικά για τις διελεύσεις και θα πρέπει να βελτιώσουμε και αυτούς τους κόμβους με μεγαλύτερη προσοχή στο διάδρομο. Και τέλος πρέπει να επενδύσουμε στο σύστημα ασφαλείας και σηματοδότησης για τους σιδηροδρόμους ο Καλβίν και το σχέδιο δράσης του θα πρέπει να υποστηριχθούν. Για μένα είναι αποφασιστικό να μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση των συστημάτων ασφαλείας και να υπάρξει συγχρονισμός όλων των προσπαθειών. Εν τέλει θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Θέλω να τονίσω ότι το σχέδιο για το διάδρομο αυτό είναι μια κοινή υποχρέωση όλων μας. Καταρχήν, το σχέδιο δράσης βασίζεται σε μια λεπτομεριακή ανάλυση των διαδρόμων, αλλά επίσης και σε μια μελέτη αγοράς πολυτροπικού χαρακτήρα. Ο, στό, ο στόχος μας είναι, θα πρέπει να είναι μέλλον να διαχειριστούμε σωστά τα ρεύματα κυκλοφορίας και να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική μεταφορών της Ευρώπης θα είναι λειτουργική. Και επίσης αυτό το οποίο τόνισα είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εμπλεκομένων που θα πρέπει να τύχουν διαβούλευση αλλά παίξουν και ρόλο στην εργασία μας. Γι' αυτό έχουμε οργανώσει φόρουμ για τους διαδρόμους της Βρυξέλλες που με τρόπο ε, σταδιακό έχει περιλάβει τα κρατημέλη μετά τους διαχειριστές υποδομών στα διάφορα για τις διάφορες μορφές μεταφορών, λιμάνια, αεροπλάνα, βαπόρια κτλ. Επίσης είχαμε ομάδες εργασίας θεματικού χαρακτήρα για τους λιμένες και τους εκπροσώπους των εμπλεκομένων περιφερειών και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε αυτές τις επαφές με στα κράτη-μέλη για όλους αυτούς οι οποίοι αναπτύσσουν τους διαδρόμους και αυτό είναι πιστεύω σωστός δρόμος που θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε και φυσικά είχαμε για τα διαμεθοριακά σχέδια επαφές σε διμερές επίπεδο. Έχω επισκεφτεί όλες τις ε, χώρες εμπλεκόμενες και σε διμερές επίπεδο και σε κοινέ συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους υπουργού έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά. Κάναμε πολλές διμερείς επαφές. Όχι μονάχα για τις διαμεθοριακές αλλά και για άλλες περιπτώσεις. Και τέλος Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών. Αυτό το ερώτημα το έθεσε και ο βουλευτής από την ε, Μάλτα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, υποδοχή μου. Με επιφυλάξατε και την πρόσκληση. Ευχαριστώ Κουρτ, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα τα ερωτήματα. Ο Μασιλιάνος Σαλίνη πρώτος. Buongiorno, grazie mille, coordinatore Ε, γεια σα είμαι συντονιστή έχω τα δύο να σα πω. Πρώτα πρώτα, Ακριβώ για το πόσο σημαντικό είναι αυτό ο διάδρομο βαλτική Αδριατική. γιατί αν αμφίβολα η προοπτική για την ανάπτυξη της Ευρώπη είναι αυτό, δηλαδή να ε, υπάρξει αυτού του είδους η σύνδεση που προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό κάνει ακριβώς και ο διάδρομος που ξεκινάει από το βορρά και καταλήγει στη χώρα μου την Ιταλία. Έχω δύο ερωτήσεις που έχουν σχέση με την εμπλοκή της χώρας μου στην υπόθεση. Πρώτα πρώτα, τι σχέση έχει η στρατηγική ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας των Άλπαιων είναι κάτι που κυριαρχεί σε αυτή την ε, περιφέρεια, σε αυτή την περιοχή της Βορειοιταλίας, εκεί όπου έχουμε αυτόν τον κόμβο για τον διάδρομο που συζητούμε. Εσείς τι συντονισμό θα κάνετε στρατηγικού χαρακτήρα όσον αφορά επομένως τη Σάλπις και από την άλλη μεριά της προσπάθειας για τον διάδρομο. Τώρα κάτι άλλο. Κάτι για τους λιμένες της Βορείου Αδριατικής. Εκεί έχουμε μια σειρά από Ιταλικούς λιμένες που ανοίγουν σε αυτό το σημαντικό κομμάτι του διαδρόμου. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο συζητηθεί πάρα πολύ στην Ιταλία και ο εμπνευστής του ήταν ο Παύλο Κώστο που το γνωρίζουμε πάρα πολύ στην Επιτροπή μας και υπάρχει αυτό το σχέδιο λοιπόν, που σχέση με το λιμένα της Βενετίας συζητήθηκε είπαμε πολύ στην Ιταλία και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτό το έργο, αυτό το σχέδιο. Θα μπορούσε να είναι μια εξέλιξη πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί αν το σκεφτούμε και σε σχέση με τη διεύρυνση του ΣΟΕΖ, τότε έχουμε ε, πραγματικά την ε, ε, δυνατότητα να αναδεχθούμε ένα σωρό εμπορεύματα τα οποία θα, θα ερχόντουσαν από κάτω προς την Ευρώπη, αλλιώς αν δεν υπήρχε αυτό το έργο, τότε θα χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Λιμπεράτσικη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, για όσο μας είπατε, ευχαριστούμε. Μας μίλησατε για αυτόν τον ε, διάδρομο που αφορά την Βαλτική και την Αδριατική. Πολύ σημαντική σημερινή συζήτηση που έχουμε απόσταση 220 χιλιόμετρα μέσα στο εδαφό μας μεταξύ των δύο διαδρόμων οι οποίοι ενώνονται κάτω στην Αυστρία. Και ο πρόεδρος μου, κύριος Καραμάρ, στην αρχή μας ανέφερε αυτά τα σημαντικά προβλήματα όσον αφορά το Αμβούργο και όπου έχουμε αυτά τα προβλήματα της συμφόρησης για την ε, κυκλοφορία εκεί. Επομένως να είναι αλληλεκτική λύση που είναι αυτός ο διάδρομος. Ή επίσης ε, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες επενδύσεις σε Σκανδιναβία, στη Γερμανία και έτσι να έχουμε ένα άλλο κομμάτι και να βοηθάει τις μεταφορές ε, και επομένως και αυτό να καλυφθεί στα πλαίσια του, του σχεδίου. Τώρα, έχουμε τη σύνδεση Ντάνς Καροβίτσε, Βαρσοβία, Ούτς, Κατοβίτσε και είπαμε ότι αυτό ξεκίνησε, έπεσε η διάσταση του 2013. Επίσης, ε, Στετίνο, Πόσναν, ένα άλλο κομμάτι. Και μετά έχουμε τη σύνδεση μέχρι την Οστράβα για τον ε, διάδρομο αυτόν που ε, έχει ξεκινήσει από, τον Ντάντσεκ και μετά διασχίζει Γερμανία και, Αύστρια, και Αυστρία. Οπότε τώρα συνεχίστε μετά προς, ε, προς νότον αυτός ο διάδρομος και σας ερωτώ κύριε Υπουργέ, κύριε Συντονιστά έχουμε το διάδρομο υπαριθμών 3 και πολύ σημαντικό σαν έργο υποδομής γιατί ε, συνδέει στην Ελβετία το Ίστατ με την Νότια Ελβετία. Συγγνώμη, Σουηδία. Και κατόπιν ε, περνάει και έχουμε τη διαδρομή της οδρομική που είναι πολύ σημαντική για μεταφορά εμπορευμάτων και ξεκινάμε η επόμενη διαδρομή από το Στετίνο μέχρι το Βρότσλαφ. Και επίσης έχουμε και την, τη σύνδεση που φτάνει μέχρι την Μπρατισλάβο. Έχω την εξή ερώτηση. Έχουμε μια σύραγγα εκεί, κάτω από το, ποτάμι Σφίνα της ε, χώρας μας. Μήκος 1600 μέτρα. Δεν είναι πολλά, όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τις μεταφορές Πολωνίας, Γερμανίας, γιατί μιλούμε για, για τα σύνορα των δύο χωρών. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μια εξαιρετικού χαρακτήρα περίπτωση. Δεν μιλάμε για κάποιον κόμβο, για κάποια ε, σύνδεση κατά ξηρά, αλλά μιλάμε για κάτι που περνά κάτω από το ποτάμι. Και το θέμα τώρα είναι τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Ε, αυτό, το, το, το, αυτή η υπόθεση του, διαδρόμου πώς εντάσσεται στο σχέδιο Γιούνκερ. Έχουμε προβλέψεις για κάποιες χρηματοδοτικές ε, ε, μεθόδους όπως τα ομόλογα έργων. Γιατί τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να καλυφθεί ένα τμήμα της υποδομής. Γιατί ε, πρόκειται για ένα τομέα όπου θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατασκευή της υποδομής με συμμετοχή Γερμανίας αλλά και Σκανδιναβίας. Ε, επίσης το, το, το, το ποσοστό της απόδοσης και της επιστροφής θα πρέπει να είναι κάτι που προχωράει γρήγορα γιατί πολλές φορές έχουμε καθυστερήσεις όσον αφορά τις ε, επενδύσεις. Οπότε θα πρέπει εδώ να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα χωρίς να επιστρατεύσουμε μεγάλο τμήμα των ε, επενδύσεων. Έχω κι άλλο ένα ερώτημα όμως. Μιλούμε για αυτό το σχέδιο που το ονομάζουμε ε, διαδρομή 3 ε, και σύνδεση διαδρομική για τα εμπορικά τρένα. Όλα αυτά δεν καλύφθηκαν, εξηρέθησαν η πολωνική κυβέρνηση ε, φταίει που ήθελε να ευνοήσει τη σύνδεση με το Δάντζεχ ή έχουμε και άλλους λόγους που δεν καλύφθηκε. Η Κλάουδια Σμιτ. έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέντεβικ πάρα πολύ για την παρουσίαση και το έργο, το έργο το οποίο χρειαστεί για να δημιουργηθεί αυτή η μελέτη. Εγώ σίγουρα υποστηρίζω τις πρωτοβουλίες οι οποίες οδηγούν σε καλύτερη σύνδεση μεταξύ των τμήματων της Ευρώπης και νομίζω ότι αυτές οι, μεταφο... συνδέσεις μεταφορών δεν είναι μονάχα συνδέσεις μεταφορικού χαρακτήρα, αλλά διηγούν σε ανάπτυξη επιχειρήσεων και οικονομική ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά. Το πρώτο μου ερώτημα είναι αν υπάρχουν κάποιες ε, εκτιμήσεις για το πώς θα επηρεάσει αυτός ο διάδρομος τις περιοχές και, την, και τις χώρες από τις οποίες περνάνε. Και επίσης για τα δύο μεγάλα τούνελ που αναφέρατε στην Αυστρία, το Σεμαρίν και το Κοαρίν τούνελ, χωρίς αυτά τα δύο σχέδια. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θα μπορέσουν να συνδεθούν στο διάδρομο. Υπάρχουν προβλήματα όμως στην Αυστρία με την προστασία του περιβάλλοντος και υπάρχουν ομάδες οι οποίες προσπαθούν να εμποδίσουν την πραγματοποίηση αυτών των σχεδίων. Και ξέρω ότι υπήρξε μεγάλη αντίδραση όταν είπε η κυρία Μπούλτς ότι δεν θα προχωρήσουν αυτά σε πρώτη φάση. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν εσεί ε, ε, μπορούσατε να κάνετε κάποια σχόλια με τη συγχρηματοδότηση αυτών των σειράγκων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια σωστή χρηματοδότηση για αυτές τις ε, υποδομές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει να έχει κάνει την γνώμη του και να την εκφράσει παρά το γεγονός ότι διαφωνώ μαζί σας. Αυτό <laughs> δεν έχει, που έχετε να κάνετε με η Αυστρία και αυτή μια γερμανική, γερμανόφωνη περιοχή. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τις οδικές μεταφορές. θα πέσει αυτού του διαδρόμου. Αναφερθήκατε στα σημεία συμφόρησης και είπατε ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ε, συμφορήσεις, στα σημεία συμφόρησης στις οδικές μεταφορές. Στην Τσεχία, στο, ανάμεσα στο Λίπιν και στο Σνιέκοβιτσα, αναφερθήκατε και, και εσείς αυτό εξάλλου, ε, υπάρχει ένα σημείο συμφόρησης γνωστό, αυτό και πάρα πολύ καιρό. Επίσης, ε, αναφερθήκατε στην ε, σύνδεση ανάμεσα στη Γέννη και στο Βενόκ. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σχεδία για αυτά τα σημεία. Ο πετατός Πώς επίσης ε, μας μίλησε για τα προγράμματα σε σχέση με την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών και τη χρηματοδότηση από το ΣΕΦ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε το ΣΕΦ και το κονδύλι της συνοχής να δώσει μια χρηματοδότηση για αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα του διαδρόμου. Σας ευχαριστούμε για την werde. Ευχαριστώ πολύ και από την πλευρά των φιλελευθέρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που ήρθατε εδώ. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα. Μιλήσατε για ε, θαλάσσιους λιμένες και εσωτερικούς λιμένες. Δεν είπατε τίποτα για εσωτερικές ε, υδάτινες οδούς. Τι ρόλο παίζουν μέσα στην, στο διάδρομο αυτό βλέπετε. Εγώ βλέπω ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά για τους ε, σιδηροδρόμους. Αλλά νομίζω ότι με τις εσωτερικές υδάτινες οδούς μπορεί κανείς να κάνει περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό το τέταρτο πακέτο για τα σιδηροδρομικά στο τεχνικό του τμήμα, σε ποιο βαθμό θα βοηθήσει τον διαδρομό σας Είπατε ότι έχετε τρία διαφορετικά συστήματα ηλεκτροδότησης. Μήπως χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη εναρμόνιση και θα ήταν πολύ χρήσιμο το τέταρτο πακέτο. Θα παραμείνω λοιπόν σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Για τις εσωτερικές ιδιαίτερες οδούς και για την ηλεκτροδότηση των γραμμών. Και εγώ θα λάβω το λόγο. 53% για το σιδηρόδρομο Καλό φαίνεται, αλλά αν βάλουμε και τα ε, τούνελ, είναι πολλά χρήματα τα οποία θα πρέπει να πάνε στα τούνελ. Δηλαδή μειώνεται ο, ο αριθμός των χιλιόμετρων που θα καλυφθούν. Βλέπω στο χάρτη να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα από την ε, ε, Λουμπιάνο στην Πρατισλάβα. Μπορεί να περάσει κανείς τώρα το υψίπεδο της Πανωνίας και εκεί θα μπορούσε να υπάρξει μια δυνατότητα διέλευσης από εκεί. Γιατί δεν έχει γίνει ηλεκτροδότηση λοιπόν ε, από εκείνη την περιοχή όταν τα τούλε χρειάζονται τουλάχιστον 10 χρόνια. Εγώ είμαι καταρχήν εναντίον των συλλάγων, αλλά αφού δεν μπορούν να γίνουν αρκετά γρήγορα, νομίζω ότι οι άλλες δυνατότητες θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητα. Και ξέρω ότι μπορεί να ενοχληθούν οι αστριακοί με αυτό που λέω, Αυτό μπορεί να συζητηθεί από τους ίδιους τους ε, Αυστριακούς, αλλά εγώ νομίζω ότι αναρωτιέμαι γιατί υπάρχουν αυτά τα προγράμματα τα οποία παίρνουν χρηματοδότηση και το ίδιο γίνεται για το Fairman Belt. Το Κόραν και το Σέμερινγκ είναι θέματα που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ καιρό στην ε, ε, Αυστρία και από τους πράσινους που έχουν κερδίσει δύο δίκες είναι περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος από την UNESCO. Το θέμα είναι αν αυτό αφορά μόνο αυτό το σιδηροδρομικό κομμάτι, του Σύνδρο του σχεδίου και υπάρχουν από τον καθηγητή Κλον Φλάχερ ε, μια πραγματογνωμοσύνη για τα θέματα αυτά που είπε ότι αυτά τα τούνελ θα είχαν παράγοντα κόστους, ωφέλειες κόστους 0,15 με 0,20. Αν φτιάξουμε λοιπόν το τούνελ της Ζέμερεγκ αυτό θα, δεν θα οδηγούσε σε τίποτα. Λοιπόν, τώρα πώς θα ελεγχθούν αυτά, δεν ξέρω τώρα αν είναι έγκυρα τα αριθμητικά στοιχεία, στα σχέδια αυτά θα πρέπει να έχει κανείς πραγματικά μια ε, βεβαιότητα. Για την ε, διατήρηση επίσης υποδομής χρειαζόμαστε 7,2 δισεκατομμύρια το χρόνο υπολογίζεται για τη διατήρηση της ε, υποδομής. Και αυτό το λέει και το γερμανικό σύστημα σχέδιο για τις μεταφορές. Αλλά το ξέρετε εσείς ως πρώην υπουργό Μεταφορών ότι αυτά είναι μονάχα επιθυμίες. Πώς λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουμε ποιες προτάσεις μπορούν να υποστηριχθούν ή όχι. Μόνο αν έχουμε γενικά διόδια σε όλη την Ευρώπη θα μπορέσει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά θα έχουμε δυσκολία με τα αυτοκίνητα των ξένων. Και σας δίνω τώρα το λόγο κύριε Μπόντεβιν. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευρία βεντάλια ερωτημάτων που αφορούν από λεπτομεριακά θέματα μέχρι στρατηγικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για το ευρύ αυτό φάσμα ερωτημάτων. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Σαλίνη με αυτό τον ε, διάδρομο κάνουμε, δημιουργούμε νέο έδαφος. Θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και την συνεκτικότητά της. Θέλουμε να εστιάσουμε στα θέματα <clears throat> μεταφορών και η θετική ιδέα για αυτό το δίκτυο είναι ότι μπορούμε να συνδέσουμε την Αδριατική με την Βαλτική και αυτό θα ανοίξει νέες δυνατότητες. Και έρχομαι στο ερώτημα που είπατε ποιε θα είναι οι συνέπειες σε μακροοικονομικό επίπεδο για τις χώρες από τις οποίες διέρχεται αυτός ο διάδομος, αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ε, ζητώ την κατανόησή σας που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τίποτα για τους, εξοχ, για τους υπεράκτιους λιμένες. Δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος που θα μπορούσε να προκύψει για ένα τέτοιο σύστημα. Θα πρέπει αυτά να τα ελέγξει για να έχει μια καλύτερη ιδέα για το οικονομικό κόστος. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ε, μελετών. Το ένα ήταν για τις τεχνικές δυνατότητες και το δεύτερο επίπεδο είναι ποια είναι τα σχέδια, σε ποια φάση θα έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική αξία. Οι μακροϊπεριφέρειες της ΑΛΠ των Άλπαιων και άλλες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γι' αυτό έχουμε και ένα πάνελ μέσα στον, στους ενδιαφερμένους για αυτό το διάδρομο, όπου υπάρχουν στη DigiMove και εκπρόσωποι της DigiRegio και αυτό έχει κάθε νόημα όταν θέλουμε να αναπτύξουμε ε, στρατηγικές μακροπεριφερειακές, οι οποίες συνδέονται με στρατηγικές μεταφορών. Ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό έχω κάπως καλύψει το ερώτημά σας. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις μεμονωμένες επιθυμίες σε ένα συνολικό πλαίσιο και εγώ φυσικά είμαι από τους υπέρμαχους των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και έχει φανεί και αυτό στην περίπτωση της Βαλτικής και αυτό προωθεί ιδιαίτερα αυτές τις στρατηγικές. Για τον κύριο Λιμπεράτσκι, ο οποίος και αυτός υπήρξε υπουργό Μεταφορών και φυσικά γνωρίζει σε βάθος τα θέματα αυτά και λεπτομεριακά. Είναι σωστό ο διάδρομος αυτός, η διάδρομη αυτή μάλλον συνδέονται. Το... Ο διάδρομος αυτός και ο διάδρομος ο, ο οποίος πηγαίνει ανατολικά δυτικά τέμνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς μέσω των διαδρόμων αυτών με την ε, διαδρομή προς το Σέσιν Σινούτσε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Το έχουμε παράλληλες λοιπόν διαδρομές είναι σημαντικό να αποφασίσουμε αν αυτό είναι η καλύτερη λύση ή αν θέλουμε να φέρουμε τις περισσότερες επενδύσεις σε ένα σύστημα το οποίο μετά μπορεί να διαφοροποιηθεί στο μέλλον. Και έχουμε για τον διάδρομο αυτό Βαλτικής Αδριατικής έχουμε εστιάσει την προσοχή αυτή στο ERTMS 5. Θέλουμε οι σιδηροδρομικές αυτές ε, ε, συνδέσεις να έχουν μια λειτουργική ε, αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές και να ακολουθούμε όμως συγχρόνως και τον κανονισμό των διευρωπαϊκών δικτύων και να βασίζεται σε αυτό. Από την πλευρά αυτή είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι και στην Πολωνία θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους λιμένες αλλά και τις πόλεις οι οποίες συνδέονται με την διαδρομή αυτή θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε την ανάπτυξή τους. Θέλω να κάνω πολύ σαφές. Έχουμε σχέδια Ανάπτυξη τα οποία τα έχουμε συνδέσει με την συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο λοιπόν προετοιμάζεται στη Γερμανία και στι άλλες χώρες πρέπει να συνδεθεί με αυτούς τους διαδρόμους και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η εθνική σχεδίαση για τους διαδρόμους συνδέεται με το σχέδιο δράση για το διάδρομο. Τα ερωτήματα τώρα για το ΕΦΣΥ. Ο κ. Ζιμπεράσκη ρώτησε κατά πόσο το, σχέδιο Γιούνκερ ε, μπορεί να ενθαρρύνει την ε, ανάπτυξη αυτών των σχεδίων. Έχουμε μια δυνατότητα να αντλήσουμε μεσοπρόθεσμα 16 δισεκατομμύρια για την, ε, το διάδρομο αυτό και ανεξάρτητα από το Ταμείο Συνοχής. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν για τα σχέδια τα οποία μπορούν να έλθουν το ταχύτερο δυνατό και τα οποία μπορούν να πάρουν μια διαφορετική χρηματοδότηση. Και επίσης, για το ερώτημα το οποίο έθεσε η κυρία Σουμίτ προηγουμένως, τα σχέδια πρόκειται φυσικά όπως σας είπα για την πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Δεύτερον, για σχέδια τα οποία ξεπερνούν το μεσοπρόθεσμο χρηματοδοτικό διάστημα και επίσης υπάρχει δυνατότητα μέσα στο ΕΦΣΥ να υπάρξουν τέτοια προγράμματα. Με την έκθεση αυτή, την λεγόμενη έκθεση CVS, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα είδος ηλιοτυπίας για τη μελλοντική ανάπτυξη των διαδρόμων αυτών που να έχει χρηματοδοτική εφικτότητα. Και με το σχέδιο Juncker έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο και ακολουθούμε ένα σωστό δρόμο. Είπατε κυρία Σμιτ ποια είναι τα οικονομικά αποτελέσματα, τα θετικά. Υπάρχει μια μελέτη του Ιδρύματος Φραουνχόφερ που υπολογίζει ποια είναι τα οικονομικά, τα μακροοικονομικά αποτελέσματα της μη δημιουργίας αυτών των διαδρόμων. Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεων εργασίας και δεν είναι το 1 προς 4 που ελέγχθη. Ο στόχος μας είναι με τη δημιουργία μιας υποδομής να έχουμε καλύτερη επιμελητία και καλύτερη σύνδεση σε ε, οικονομικό επίπεδο που θα οδηγήσουν καιρό σε 10 εκατομμύρια θέσει εργασία. Γιατί κυρία Σέχνάλογα, φυσικά και οι οδικοί άξονες έχουν μια μεγάλη σημασία αλλά στο μεγάλο πακέτο το οποίο προβλέπεται για κάθε χώρα μόνο 10% της χρηματοδότησης προβλέπεται για τους δρόμους. Πρέπει να έχουν λοιπόν μεγάλη προτεραιότητα, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι συνδεδρομικές συνδέσεις θα πρέπει να πάρουν πολύ μεγαλύτερη ε, υποστήριξη. Φόβαμαι κυρία Μάισερ θα σας απογοητεύσω δεν παίζουν μεγάλο ρόλο οι εσωτερικές υδάτινες οδοί, αλλά μόνο στους εγκάρσιους ε, διαδρόμους και θα προσπαθήσουμε με τους θερματικούς σταθμούς να εξασφαλίσουμε καλύτερη ολοκλήρωση με τον διάδρομο μας και για το τέταρτο πακέτο για τις, ε, τα συνδρομικά πιστεύω πράγματι ότι είναι πάρα πολύ θετικό, μπορεί να βελτιώσει τις ευκαιρίες που έχουμε να έχουμε καλύτερες αναπτύξεις υποδομών. και το τελευταίο ερώτημα τώρα του κυρίου Κράμερ. Λέτε ότι 13% των κονδυλίων πηγαίνουν στα, στις, στις και αυτά είναι φυσικά πολύ δάπανα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Εδώ έχουμε μια, ένα εσωτερικό κανονισμό κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σχέδιο δράσης έξω από του τις διαδρομές αυτές που έχουν προβλεφθεί. Έχουμε την ε, διαδρομή από το Γκράτ στο Κλάγκενφουρτ που πρέπει να την ακολουθήσουμε. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό όμως για τους διαδρόμους έχουμε κάνει μελέτες και έχουμε μια μελέτη για τον περίγυρο των, των μεταφορικών αυτών διαδρόμων. Τι θα γίνει αν λειτουργήσουν ή αν δεν λειτουργήσουν λοιπόν αυτοί οι διάδρομοι. Επομένως, όταν δεν λειτουργήσει η μεταφορά με σιδηρόδρομο γιατί δεν είναι ελκυστική. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει μεταφορά της κίνησης στο δρόμο, στις οδικούς άξονες, Αυτό είναι κίνδυνος και εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε όσο και περισσότερο να είναι οι μεταφορές στο σιδηρόδρομο στο διάδρομο μας. Ευχαριστώ πολύ. vielen Dank. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Σας ευχόμαστε όλα καλά να πάνε και σίγουρα σε ένα χρόνο θα ξαναβρεθούμε και θα δούμε και πάλι πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπόδεφερ και ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt Visa-Paket. Ερχόμαστε τώρα στις ε, θεωρήσεις περιοδίας. Είναι ο κύριος Ουέ εισηγητής και του δίνω αμέσως και αδιαλείπτως το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό είναι αντιδραστήρας. Θα περιμένω λίγα λεπτάκια για να είμαι σίγουρος ότι όλοι μπορούν να βάλουν τα ακουστικά. Έχουμε δύο σημεία στη διάταξη. Προτείνω να τα δούμε από κοινού. Θα ήθελα λοιπόν να Σα δώσω τι λεπτομέρειε εσεί θα αποφασίσετε, Πρόεδρε, αν ε, πρέπει να γίνει κοινή συζήτηση ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν να τα συζητήσουμε από κοινού. Ναι, τι λέτε. Ναι, ναι, ναι, έτσι ναι. ε, το είχαμε προγραμματίσει. Συνάδελφοι. Τι θα λέγατε αν μπορούσατε να γυρίσετε στην εκλογική σας περιφέρεια και να ανακοινώσετε το εξής. Έχουμε ένα πακέτο, μία απλή τροποποίηση νομοθετικού πακέτου εφαρμοστέα για την επόμενη πενταετία όπου θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 1,3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Τι λέτε έκανε κάποιου υπολογισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση και προκύπτει 130 δι σε έσοδα μπορούν να παραχθούν την επόμενη πενταετία. Χωρίς ιδιαίτερη επένδυση, χωρίς να διοικητεύσουμε εκεί κονδύλια. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα περίπλοκο και παροχημένο νομοθέτημα για τις θεωρήσεις ε, και να το τροποποιήσουμε. Νομίζω ότι θα σας χειροκροτούσαν σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια και θα επικροτούσαν τη δράση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν ανακοινώνουν τόσο καλά νέα. Ξέρω φυσικά ότι ε, ε, μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για, ε, για το χώρο Σέγγεν, αλλά στον χώρο Σαγγέν μιλάμε για πρόσθετα έσοδα και για πρόσθετε θέσει εργασία και εξάλλου αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά χάρη στι αλλαγέ που προτείνονται μέσα σε αυτά σε αυτές τις δύο νομοθετικές ε, ρυθμίσεις. Αυτό θα μας απασχολήσουμε με τις δύο Από το Μάιο ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα. Ε, έχω κάνει πάρα πολλές ε, συναντήσεις με τους συναδέλφους, με τους κοιόδες. Και μέχρι την Κίνα φτάσαμε για να ακούσουμε και ε, τους εμπειρογνώμονες και να συλλέξουμε πληροφορίες. Μπορώ να σας πω ότι για τον τουρισμό και τις μεταφορές, ε, τα δεξοχήν θέματα αρμοδότητας της Επιτροπής μας ε, είναι κύριε σημασία να προωθήσουμε αυτούς τους δύο φακέλους στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να δούμε το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες το φθινόπωρο θα καταθέσω ε, την έκθεση της Επιτροπής Τραν μετά από την υποβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας παραπέμψω καταρχάς την έκθεση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 για τις θεωρήσεις, τις διαδικασίες, τα οικονομικά ωφέλη αυτών των συστημάτων και όπως έλεγε στην αρχή της παρέμβασής μου και τι λέει αυτή η μελέτη λέει πως αν δείτε τους κανόνες Σέγγεν που είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εφαρμόζονται και με ιδιαίτερη αυστηρότητα, εάν εξετάσετε την εφαρμογή τους και δείτε την κατάσταση τους προς τον ανταγωνισμό, έχουμε μια κατάσταση επιζήμια. Έχουμε απολέσει περίπου 6,6 εκατομμύρια τουρίστες εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η απώλεια. Για τουρίστες από την Βραζιλία, από την Ινδία, την Κίνα, τη Ρωσία, από τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να έρθουν, που είναι φερέγγοι, που είναι εύποροι και άρα θα κατανάλωναν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους χάσαμε ε, λόγω ε, του συστήματος ε, έκτος θεωρήσεων που τους αποτρέπει. Σήμερα το πρωί συναντήθηκα ε, με τον έναν από τους διευθυντές μιας μεγάλης εξοδοχειακής αλυσίδας από τη ΣΥΠΑ και μου έλεγε ότι από για μας καλό είναι άμα συνεχίσετε έτσι και άμα δεν καταλαβαίνετε εδώ στην Ευρώπη πόσο πιο ευέλικτοι πρέπει να είναι οι κανόνες για τις θεωρήσεις ε, τόσο το καλύτερο για μας γιατί θα έχουμε περισσότερους τουρίστες. Ε, στο παρελθόν ε, η Ευρώπη ε, περηφανευόταν γιατί ήταν ο πρωταρχικός ο προορισμός. Τώρα όμως είμαστε ρογές σε σχέση με την Αυστραλία, με τη ΣΥΠΑ, με την Νότια Αφρική. Αλλά θα ήταν να προσελκύσουμε λοιπόν περισσότερους τουρίστες από τις τρίτες χώρες και έχουμε τρεις, δύο διαφορετικές προτάσεις, δύο πακέτα προτάσεων αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα, αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων που είναι αυτή τη στιγμή ενισχύ και μιλάμε και για ένα νέο είδος θεώρηση, την Touring Visa, θεώρηση περιοδίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόκειται για ε, βροχέ παραμονέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκθεση θεωρήσεων για τέτοιε βροχέ παραμονέ. Ε, απλούστευση λοιπόν ε, και συντόμευση της διαδικασίας, μείωση της γραφειοκρατία και του κόστος και κάτι άλλο που επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά αξίζει να το τονίζουμε επανειλημμένα και για τις άλλες επιτροπές και το τονίζω γιατί και άλλοι θα ασχοληθούν με αυτό διότι δεν υπάρχουν μόνο τα οικονομικά ζητήματα, υπάρχει η πτυχή της ασφάλειας. Εξυπακούεται ότι τα θέματα ασφάλειας θα πρέπει να συμπολογιστούν και πάλι όμως σας λέω συνάδελφοι, 6,6 εκατομμύρια τουρίστες χάσαμε, εύπορους τουρίστες που ε, θα κατανάλωναν πάρα πολύ εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσοι από αυτά τα 6,6 εκατομμύρια θα ήταν δυνάμει τρομοκράτες, πιστεύετε εσείς. Ε, ακούω διάφορους να προτάσουν αυτό το επιχείρημα εδώ στο Κοινοβούλιο και λόγω των τελευταίων περιστατικών ε, συνέχεια με λαμβάνουν ε, αυτή την εποχή και λένε όχι πρέπει να φτιάξουμε φράκτες και να αποτρέπουμε τους ανθρώπους όχι να διευκολύνουμε ε, την είσοδο πολιτών τρίτων χώρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όμως να αποτιμήσουμε και το κίνδυνο. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα τα δύο ζητήματα, το ζήτημα των θεωρήσεων και το μεταναστευτικό ζήτημα, είναι δύο εντελώς διακριτά ζητήματα. Ο τρομοκράτης ποτέ δεν πάει να καταθέσει αίτηση στη, για θεώρηση άμα θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πιστέψτε με, αλλά όπως ε, ε, σας είπα υπάρχουν οι Κινέζοι πολίτες, επενδυτές δεν μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη και θα μπορούσαν, θα είχαν κάθε ενδιαφέρον να έρθουν να διερευνήσουν τι επαγγελματικέ ευκαιρίε εδώ στην Ευρώπη και εμεί τι κάναμε, τους εμποδίσαμε. Ε, θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω όπως για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τα έχω πει και με συναδέλφου με του οποίου μιλήσαμε τις περασμένε εβδομάδε και συμφωνήσαμε να υποστηρίξουμε τι προτάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω λοιπόν για του υπολείπους να πω ότι πρέπει η Επιτροπή Μεταφορών να προωθήσει αυτό το, αυτή την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπω και η δια, ε, πολιτική ομάδα διακομματική συγγνώμη ομάδα, όπου ε, συζητήθηκε το θέμα και υπάρχει υποστήριξη για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ήθελα επίσης να αναφέρω τις απόψεις ε, ε συλλογικών οργανισμών ε, στην Ευρώπη που ασχολούνται με τέτοια είδη θεωρήσεων, καλλιτεχνικούς οργανισμούς, παγκόσμιους οργανισμούς τουρισμού, ξενοδοχεία, ε, θίαση, θεατρική, ε, καλλιτεχνικά, ε, καλλιτεχνικές ενός καλλιτεχνών. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι υπάρχει γενικότερη υποστήριξη, θα ήθελα όμως τώρα, επειδή θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε μέχρι το φθινόπωρο, να ασχοληθώ μόνο με κάποια κεντρικά σημεία επεξεργασία των θεωρήσεων και προθεσμίες ε, για την έκδοση θεωρήσεων. Θέλουμε να συντομεύσουμε αυτές τις προθεσμίες. Για την υποβολή αίτησης ε, θα ε, είναι δυνατόν να υποβάλλετε την αίτησή σας σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος εάν δεν εκπροσωπείτε η εν λόγω χώρα με προξενία στη δική σας χώρα. Όταν μιλάμε για μεγάλε τεράστιε επιχειρήσει. με πολύ μεγάλο τζίρο. Κινέζικε επιχειρήσει. δεν έχουν απαραίτητα την έδρα του στο Πεκίνο, Σανχάι. Μπορεί να έχουν την έδρα του σε χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά ε, αλλά θα θέλουν να, ε, για τους υπαλλήλους παραδείγματος χάρη να υποβάλουν την αίτηση για θεώρηση. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και να κάνουν διαπραγματεύσεις με το ισχύον σύστημα τι σημαίνει στην πράξη. Πρέπει να πάνε στο Πεκίνο Σανχάη, πρέπει ολόκληρη τη μέρα δηλαδή να ταξιδεύουν, να διανυκτερεύσουν εκεί πέρα, ούτω ώστε να μπορέσουν ε, να υποβάλουν την αίτηση σε ένα προξενείο Σέγγεν. Είναι μακροσκελέστατη η διαδικασία και είναι αναξιοπρεπές για να σας πω την αλήθεια διότι περιπλέκει ε, τη διαδικασία. Εμείς αν είχαμε αντίστοιχα προβλήματα θα λέγαμε όχι ευχαριστώ δεν θα πάρω. Είναι τόσο περίπλοκη διαδικασία λοιπόν που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη διαδικασία, αποφάσισαν να μην ζητήσουν θεώρηση, να μην έρθουν στην Ευρώπη και κάνανε άλλο επενδύσεις. Και το ίδιο με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ε, με θειάσους, ε. όλοι το αποφεύγουν λόγω της προπλοκότητας της διαδικασίας. Επίσης υπάρχει το ζήτημα το, της θεώρησης των πολλαπλών εισόδων και πέρα από την προθεσμία <clears throat> χρειαζόμαστε και απλούστερα έντυπα τα οποία θα μπορεί να καταθέτει κάποιος επιγραμμικά. Ε, η προθεσμία θα πρέπει να είναι κατά το όριο 15 ημέρες ε, και ε, κυρίως όταν μιλάμε για θεωρήσεις βραχίας παραμονής. Αυτές είναι οι βασικές προτάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζήτησα με ειδικού ε, από τον κόσμο των επιχειρήσεων, από τους εμπόρους και από πλευράς τους ε, ε, έχω κάποιες προτάσεις απλούστευσης για τους ναυτικούς παραδείγματος χάρη ή για τους tour operators. Εκείνοι μου προτείνουν συγκεκριμένες απλούστευσεις. Θα σας δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα. ας πάρουμε τα παράδειγμα των ΗΠΑ. Υπάρχει μεγάλη έξεση στον κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών, περισσότερο από ό,τι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ε, εισαγάγει το σύστημα μιας δεκαετού θεώρηση πολλαπλών εισόδων. Εμεί ούτε καν έχουμε εξετάσει το ενδεχόμενο. Μα γιατί όχι. Δεν μπορεί κάποιο να ισχυρίζεται ότι οφείλεται αυτό στον κίνδυνο τρομοκρατική ενέργεια. Τι να πούνε και στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά τότε. Εμείς ε, ε, στην εντολή μας έχουμε και τα ζητήματα τουρισμού πέρα από τις μεταφορές, οπότε είναι καθήκον μας ε, να υποβάλουμε μια πρόταση. Αν ναι, για το σύστημα πληροφόρησης για τις θεωρήσεις, το ΒΙΣ, θα πρέπει να φροντίσουμε, να μερμηνήσουμε τους ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα υποβολής αιτήσεις για δεκαετή θεώρηση πολλαπλών εισόδων. Και όπως σας είπα νωρίτερα, θα ήταν πολύ καλή ιδέα να φροντίσουμε ιδιαίτερε ειδικέ κατηγορίες όπως η ναυτική παραδείγματο χάρη για να μπορέσουμε στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να καταθέσουν ε, ε, μία αίτηση που θα ισχύει για ολόκληρο το χώρο Σέγγεν αυτή είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Τι θα κάνουμε με τους αερολιμένους παραδείγματος χάρη, πώς θα έχουμε ε, περισσότερες απευθείας πτήσεις ε, για περισσότερους αερολιμένες, ε, πώς γίνεται να έχουμε στα σημεία διέλευσης των συνόρων επιπρόσθετες δυνατότητες για τις θεωρήσεις για την Κίνα παραδείγματος χάρη Κίνα, μάλλον, ε, υπάρχει δυνατότητα σε ε, συνοριακούς σταθμούς με ιδιαίτερα πλουστευμένες ε, διαδικασίες να προσδίδεται κάποιος την έκθεση θεώρηση. Εμείς γιατί όχι και εμείς θεωρούμαστε καλύτερος ταξιδιωτικός προορισμός από την Κίνα. Για την αναφέρουση του κώδικα θεωρήσεων είδατε τις προτάσεις μου. Εγώ βασίζομαι για τις προτάσεις στις συζητήσεις που είχαμε με εμπλεκόμενου εμπλεκόμενους και ε, από τις συσκέψεις που είχαμε με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Α, ναι, και να πω για κάτι άλλο, για αυτή την ε, θεώρηση σέγγενε της περιοδίας, όπως ονομάζεται Touring Vision, είναι καινούριο το σύστημα και θα εφαρμόζεται σε ειδικούς τρίτων χωρών που έρχονται για περίοδο άνω των 90 ημερών, αλλά μέχρι ένα χρόνο και θέλουν να περιοδεύουν, να πηγαίνουν ε, σε διάφορες χώρες. Ε, ε, δηλαδή, δεν θα περάσουν πάνω από 90 ημέρες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως θέλουν στην επικράτεια της Ένωσης γενικότερα να μείνουν για μακρύτερο χρονικό διάστημα, όχι τρεις ημέρες, θα πρόκειται για τους καλλιτέχνες φυσικά, για επιχειρηματίες, για όσους διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, Θέλουν λοιπόν μια τέτοια θεώρηση. Να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται. Τώρα θα πρέπει να φύγουν την τελευταία ημέρα των 90 ημερών, να βγουν από το Σέγγεν και να παραμείνουν 90 ημέρες, ε, ημέρες συγγνώμη, εκτός Σέγγεν και να ξαναμπούν. Είναι ε, αποτρόπαιο το σύστημα. Θα πρέπει να αλλάξει και ε, θα συζητούσα να υποστηρίξετε αυτές τις προτάσεις μέσω αυτό του Σεπτεμβρίου μπορείτε να καταθέσετε τροπολόγια και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ. Η Κλάουδε Μοντέρο Αγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις ε, παρατηρήσεις που μας έδωσε και θέλω ευχαριστώ τον κύριο Ιστοβάνη για το πολύ όμορφο έγγραφο που μας παρουσίασε και που έχει δημιουργήσει πολλές προσδοκίες στον τομέα του τουρισμού. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες για αύξηση της απασχόλησης και στον τουρισμό και αυτό πρέπει να αποτελέσει μια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι δράσεις θα πρέπει να ενισχυθούν και ιδιαίτερα αυτές οι οποίες βασίζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο περιοριστικό τμήμα του κόσμου σε ό,τι αφορά τις ε, θεωρήσεις περιοδίας. Επομένως πρέπει να έχουμε σαφέστερους κανόνες, απλούστερους κανόνες, πιο σύγχρονους κανόνες οι οποίοι θα είναι εναρμονισμένη στο χώρο του Σέγγεν. Μεγαλύτερη λοιπόν αλληλεγγύη και μικρότερη πολυπλοκότητα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλους περαιτέρω τουρίστες. Είναι μια στρατηγική λοιπόν η οποία έχει μεγάλη σημασία για μας ως Ευρώπη γιατί μπορούμε να προσελκύσουμε τουρίστες από περιοχές όπως η Ρωσία, τους Κινέζους που ναι, την Ινδία, την Μέση Ανατολή. Να μπορέσουμε λοιπόν να προσελκύσουμε όλους αυτούς τους τουρίστες στην Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι τουρίστες όχι μόνο αυξάνουν την εσωτερική ζήτηση, αλλά αυξάνουν και την ε, ανάπτυξη σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και περιφέρειες. Έχουν λοιπόν άμεση και έμεση επίπτωση στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο αυτό το πακέτο θα πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή μας που είναι αρμόδια για τον τουρισμό γιατί εμείς είμαστε η αρμόδια επιτροπή για τα θέματα τα οποία συνδέονται έμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό και εδώ θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση της διάστασης του τουρισμού. Λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να συζητούμε το θέμα της ιστοσελίδας Schengen που θα ήταν και ένας καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια για τις αιτήσει για τις ε, ε, θεωρήσεις περιοδίας και θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στους τουρίστες, τους δυνητικούς τουρίστες. Υπάρχει το Schengen Info, αυτή η ιστοσελίδα. Θα ήταν καλύτερα όμως να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση με ιστοσελίδες οι οποίες να είναι εκ των άνω προς τα κάτω χωρίς να υπάρξει μια επικάλυψη και να διαφοροποιούνται επιγραμμικά σύμφωνα με τις ανάγκες του τουρίστα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη διακριτική ευχέρεια στα προξενία, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες, διαφορετική εποχικότητα και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε αυτήν την ιστοσελίδα Schengen όπου θα υπάρχει ένας κατάλογος με τις διάφορες καταστάσεις και τις διάφορες πληροφορίες που χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τις πολλαπλές εισόδους έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι σαφές για όλους. Τα κράτη-μέλη αποφεύγουν να εκδίδουν τέτοιου είδους θεωρήσεις και ίσως εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια πρόταση από την Κομισιόν η οποία να λάβει υπόψη αυτό το πρόβλημα. Συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Ιστεβάν για τις πολλαπλές θεωρήσεις εισόδου. Θεωρώ ότι τα πρακτικά αποτελέσματα μπορεί να μην είναι τα επιθυμητά. Γι' αυτό θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εκφέρουν τη γνώμη τους και να παρουσιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό για να μπαίνουν και να βγαίνουν πολλαπλώς οι τουρίστες. Σε ό,τι αφορά για την λεγόμενη περιοδευτική θεώρηση, διότι αυτό είναι το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό της ε, θεώρησης περιοδίας είναι μια πρόταση καινοτόμου χαρακτήρα θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθεί στην πολιτική θεωρήσεών μας και θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μας μπορεί να ευνοήσει την οικονομική δραστηριότητα σε αυτό το τομέα ο οποίος είναι τόσο κρίσιμος όπως είναι ο τουρισμός αλλά θα επηρεάσει και άλλες συναφείς δραστηριότητες όπως είναι ο τομέας των μεταφορών και της εστίασης. Έχουμε λοιπόν τις περιπτώσεις όχι μονάχα και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Καναδά από όπου μπορούμε να αντλήσουμε βελτιότερες πρακτικές. Υπάρχει το Startup Visa που έχει δημιουργηθεί για να προσελκύσει επιχειρηματίες στον Καναδά. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια πολιτική για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και στον Καναδά υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το θέμα αυτό, πάντα διατηρώντας τα απαραίτητα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, ώστε να έχουμε μια κατάσταση που προσαρμόζεται στην ε, ανάγκη ειδικών κατηγοριών όπως είναι οι καλλιτέχνες, οι αθλητές, οι φοιτητές, οι ερευνητές. Όλοι αυτοί που πρέπει να μείνουν πάνω από 30 μέρες και έχουν τη δυνατότητα και έχουν την ανάγκη να πάνε σε διάφορα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα. Ο κύριο Πρόεδρος θέλει να με διακόψει ενώ δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Πρέπει να αναλύσουμε λοιπόν όλε αυτέ τις δυνατότητε οι οποίε έχουν να κάνουν με τι προξενικέ θεωρήσει και επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, ο, επειδή μιλήσατε για τα ποδήλατα και την περιοδία που μπορεί να γίνει με τα ποδήλατα, να τονίσω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία να προωθηθεί 44 δισεκατομμύρια ευρώ δίνει στον τουρισμό γιατί ο κάθε τουρίστας είναι δυνητικός ποδηλάτης και ο κάθε ποδηλάτης είναι δυνητικός τουρίστας. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει ο τρόπος για να αυξήσουμε την κίνηση των ποδηλατών τουριστών. Και θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν θα μπορέσουν να, να μεταφερθούν σε τροπολογίες που θα παρουσιάσω εν ευθέτω χρόνο. Ακολουθώντας τη συζήτηση μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Αλλά δεν μπορεί τώρα ο να μιλάει 10 λεπτά. Δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε το, την ημερησία διάταξή μας. Ο Ντάνιελ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο και με τίποτα στα 10 λεπτά. Ευχαριστούμε τον ε, εισηγητή πάρα πολύ θετικό το, το πακέτο που προτάσαμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν τόσο ώστε να μπορέσουμε να, να τα ελκύσουμε και από τι επενδύσει και υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα, υπάρχουν και θέματα ασφαλείας γιατί μιλάμε τώρα και για οικονομικούς μετανάστε και για πρόσφυγες. Αυτή η θεώρηση περιοδία είναι ένα πρόβλημα έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να παρακάμψει το σύστημα και πάρα πολύ ωραία τα είπε ο εισηγητής γιατί έτσι αποθαρρύνονται κάποιοι ε, επισκέπτες. Δεν μπορούμε πάντως να παραμελήσουμε τον παράγοντα ασφάλεια, άρα χρειάζεται να υπάρξει συντονισμός με τους υπάρχοντες μηχανισμούς ασφαλείας στην Ένωση, να έχουμε το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών όπως το ΣΥΣ και το ΒΙΣ. Επίσης ένα σύστημα ε, όπου να μπορούν ε, να υποβάλουν αίτηση οι οι πολίτε των κρατών μελών και θα πρέπει επίση οι έλεγχοι να γίνονται για οποιονδήποτε υποβάλλει αίτηση, να είμαστε προσεκτικοί, να μην ε, υποβαθμίσουν του ελέγχου για κανέναν. Γιατί έτσι έχουμε παραθυράκι στο σύστημα επίση. Είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθεί το σύστημα των ευφυών συνόρων όσον τον τον κώδικα θεωρήσεων. Είναι και αυτό μια πρακτική ε, πρωτοβουλία ιδίως αυτό το website με, ε, με ενημέρωση, με ηλεκτρονικά έντυπα, ε, επίσης για τη συνέντευξη, πολύ σημαντικό. Όμως προβληματίζομαι σε σχέση με όσα πρότεινε η Λίμπε και η Κομισιόν. Να σας πω ποιες είναι οι επιφυλάξεις μου. Εκεί που λέγεται κατάργηση της ανάγκης υποβολής εγγράφων, ε, να αποδεικνύει ότι έχει μέσα επιβίωσης ο ε, ετών, και τι θα γίνει επίσης με την πρόθεση παραμονής ή όχι ε, του τακτικού ταξιδιώτη. Αυτό έχει σημασία για τους ε, παράνομους μετανάστες. Επίσης θα πρέπει να δούμε προσεκτικά τι θεωρήσει χορηγούμε σε όποιον θέλει να έρθει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να καλύψουμε τα παραθυράκια. Ποιο δηλαδή ισχύει ότι είναι τουρίστα. Δεν είναι θέμα ασφάλεια και ε, τρομοκρατών. Θα ε, ε, δούμε τι είναι θέμα παράνομων μεταναστών. Και έχουμε για τι ανθρωπιστικέ θεωρήσει. Θα πρέπει να πάνε σε κάποιο άλλο μέσο πολιτική και με ανησυχεί. Το ότι αν έχουμε χωριστή ρύθμιση τότε πάρα πολλοί θέλουν να διασχίσουν την ε, Μεσόγειο. Θα είναι σαν να τους λέμε καλώς τους. Οπότε, συμφωνώ επί της αρχής με αυτή τη δέσμη μέτρων, συμφωνώ και με τον εισηγητή, αλλά θα πρέπει να ξεσορροπήσουμε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις με την ασφάλεια. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η πρώτη τελευταία απόψεων, οπότε και εγώ θα είμαι σύντομη και θα προσπαθήσουμε να αυτή την ε, κοινή τοποθέτηση, βεβαίω και άλλαξαν οι καιροί. Και οι εκθέσει των επιπτώσεων είναι μπροστά μα για την καινούργια οικονομική κατάσταση, για την σχέση της Ένωσης με τον κόσμο. Αυτά μας υποχρεώνουν να αλλάξουμε γνώμη και απόψη σε σχέση με τις ε, θεωρήσεις. Βεβαίω και συμφωνούμε θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία, να διευκολύνουμε αυτούς που θέλουν να υποβάλουν αίτηση από το ίντερνετ, επομένως να έχουμε ένα σύστημα, μια μέθοδο ευέλικτη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υποδεχθούμε ε, κόσμο από τις τρίτες χώρες. Τώρα για τις οικονομικές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο ζητήματα εμπορικά, Άρα θα πρέπει να καλύψουμε τις ε, συμφωνίες που τώρα βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τρίτες χώρες και αυτές που θα διαπραγματευτούμε με τις τρίτες χώρες. Να είμαστε συνεπείς επομένως ε, αφενός ε, με τη ρύθμιση των θεωρήσεων και από την άλλη μεριά αυτό να συνάδει προς τις συμφωνίες. Τώρα, να δούμε αν χρειάζεται μία τρόπο, αν κάποια αλλαγή στο σύστημα ε, πρόκειται να μας δημιουργήσει πρόβλημα ασφαλείας. Το έχουμε δει αυτό και σε άλλες συζητήσεις. Βεβαίω δεν μπορούμε να υψώσουμε τύχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δυσκολέψουμε την είσοδο εκείνων οι οποίοι εξάλλου βοηθάνε στην οικονομική ανάπτυξη. Τώρα όσον αφορά τον τουρισμό, Έχει και τώρα τους τουρίστες, όμως θα πρέπει να καλυφθεί και αυτό αλλιώς. Γιατί εδώ πέρα καλύπτονται αυτοί που θέλουν να λάβουν βίζα. Όμως είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορούμε να, τα, να κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζονται. Τα είπαμε το πρώτο με τον Λουξεμβουργό Υπουργό. Έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για τις μεταφορές. Οπότε και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολη τη μεταφορά των ε, πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ούτω ώστε να εντάσσονται πιο εύκολα οι άνθρωποι στις τρίτες χώρες. χώρες. Επομένως εδώ δεν είναι μόνο θέμα διαβούλευσης, είναι θέμα και του πόσο συνεπείς θα είμαστε με τα υπόλοιπα θέματα που μας απασχολούν στο Κοινοβούλιο. Άρα θα πρέπει σφαιρικά να δούμε τα ζητήματα των θεωρήσεων ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παράλληλα και στα υπόλοιπα ζητήματα και πέραν της Επιτροπής των Μεταφορών και στις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Οπότε, εγώ θα προσπαθήσω να κατεβάσω κάποιες τροπολογίες ούτω ώστε να δούμε σφαιρικά το ζήτημα των θεωρήσεων. Δεν είναι θέμα το αν έχουμε βίζα για 90 μέρες και μετά 120 μέρες και μετά το κοστίζει αλφα πόσο και τι θα κάνουν. Αυτά πρόεδρε. Η Κλάουτ θα παρέλθει καλά και και άλλους δύο. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Η Κλάουδια πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Ισηγητά, κύριε Ιστβάν, αγαπητέ Ιστβάν. Σε ευχαριστώ για την έκθεση, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μέσα στο τωρινό πλαίσιο του τομέα του τουρισμού, που είναι ο τρίτος οικονομικό ε, κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά το τμήμα του ΑΕΠ που καταλαμβάνει. Άκουσα με προσοχή αυτά που ελέγχθησα στη συζήτηση και αυτά που είπε ο υπάρχει μια διαδικασία για τη διακόνηση της παροχής θεωρήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό μπορεί να οδηγήσει και ε, κέρδη από 500 εκατομμύρια ως 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τον μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα για τις θεωρήσεις. Αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Υποστηρίζω λοιπόν την γενική προσέγγιση του εισηγητή με τις διαδικασίες για την αίτηση και την ε, ε, παραλαβή των θεωρήσεων που πρέπει να είναι αντικειμενικές. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσελκύσουμε και τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα, την ε, Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία, την Ουκρανία. Πρόκειται για πληθυσμούς που έχουν μια σημαντική οικονομική δυνατότητα και μπορούν να αδειάσουν το θυλάκιό τους στις ευρωπαϊκές χώρες. Υποστήριζω λοιπόν και την απλοποίηση των αιτήσεων, ιδίως για αυτούς που είναι ήδη ε, εγγεγραμμένη στο σύστημα VES, Visa Information System. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και εξάλλου οι ετούντες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να παίρνουν τις θεωρήσεις αυτές. Και επίσης θα πρέπει να, διατηρήσουμε συγκεκριμένες ε, ε, αρχές και κριτήρια. Θα πρέπει να είναι σαφή τα κριτήρια για να μπορεί να θεωρηθεί μια επιχείρηση, ένας φορέας ότι είναι αξιόπιστος. Δεν πρέπει να υπάρχουν υποκειμενικές ή μη εναρμονισμένες κρίσεις από τα προξενία των κρατών μελών. Χρειάζεται ένα σωστός ευρωπαϊκός ορισμός που θα επιτρέψει και στα κράτη-μέλη να δράσουν όπως πρέπει. Το κόστος των θεωρήσεων αποτελεί επίσης ένα πρόβλημα, δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουμε επί τη βάση του κόστου τους δυνητικούς ετούμντες. Το κόστο αυτό θα πρέπει να είναι όσο να τον χαμηλότερο. Και μια τελευταία ιδέα που θέλω να σας υποβάλω, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, ανάλυση αντικτύπου για τη μεταρρύθμιση του κώδικα των θεωρήσεων. Μια τέτοια μελέτη όμως που είναι καθυστερήσει διαδικασία. Θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για τα κριτήρια της μελέτης αντικτύπου και οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως χρονοτριβικό εργαλείο για τις προτάσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Μάια Κίλενεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήρθα να σε ευχαριστούμε. Εσένα και το επιτελείο σου. Για την αξιόλογη δουλειά που ολοκληρώσατε. Θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε μια πολιτική θεωρήσεων που να μας δίνει τη δυνατότητα να ε, βγούμε κερδισμένοι από τον τουρισμό και η αφετηρία να είναι το τι κάνουμε με τους ε, ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, όχι, να μην θεωρούμε ότι είναι εγκληματίες. Αλλά πάντως δεν είναι ένοχοι. Δεν μπορούμε να κλειδώσουμε τα σύνορα, ούτε να επιβάλλουμε κάποιες προϋποθέσεις που θα αποθαρρύνουν τον κόσμο να έρχεται στην Ευρώπη. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τι γίνεται στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη ΣΥΠΑ, προσπαθούν να αποκλείσουν μετανάστευση από την Ασία. Πολλαπλέ θεωρήσει επομένω. Είπαμε ότι δεν τι θέλουν. Ξέρουμε όλοι πόσο αυστηροί είναι οι Αμερικανοί τόσα χρόνια. Προχωρούμε προσοχή. Δεν φτιάζονται όσοι ανθρώπου θέλουν να μπουν στη χώρα του. Εάν εμεί επομένω ε, ήμασταν αυστηροί στην πολιτική μα και αν είμαστε αυστηροί με του φοροφυγάδε αυτοί κλέβουν τα λεφτά τη Ένωση. Αν ήμασταν λίγο αυστηροί, θα είχαμε τόσα λεφτά, δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Danke sehr. Jetzt du Bravka Suiza. Die Kirche Suiza. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα Να ευχαριστήσω την Τρέστον για τη δουλειά που έκανε. Ξέρετε, είμαι από την Κροατία και είναι λίγο συστηματικά φορτισμένο το ζήτημα για μένα. Ε, μετά από δύο χρόνια προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, ε, ανήκουμε στο Σέγγεν. χρειάζεται να ζητούμε ξεχωριστή θεώρηση για τη ΣΥΠΑ, παραδείγματος χάρη, αλλά αυτό δεν ισχύει για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Τέλο πάντων, ας μην παραφέρνουμε τώρα από συναισθηματισμούς. Χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση, διότι υπάρχει η οικονομική πτυχή και η πτυχή της ασφάλειας. Θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ στην οικονομική πτυχή. Ο τουρισμός είναι βασική πλουτοπαραγωγική δραστηριότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τουρισμός τρίτος σειράς προς την δημιουργία ε, του εισοδήματος και... Οι τουρίστες από την Κίνα, από την Ινδία και γενικότερα από την Άπο Ανατολή μπορούν να προσφέρουν μεγάλα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας είπε και ο εισηγητής. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε ειδικέ κατηγορίες για τους ναυτικούς, για όσους ε, εργάζονται σε μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις και ούτω καθεξής. Αυτό το ποσό που αυτό αυτό το αριθμό των 6,6 εκατομμυρίων είναι κάτι που θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε, διότι ε, όταν μιλάμε για τόσες νέες θέσεις εργασίας, τις χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. για την, το μεταναστευτικό ζήτημα ε, εξεπακούεται θα πρέπει να βελτιώσουμε το πακέτο για τα ευφυή σύνορα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να φροντίσουμε ε, το θέμα των θεωρήσεων. Θα σας βοηθήσουμε με τις τροπολογίες μας, ώστε να εμπλουτίσετε την έκθεσή σας. Σας ευχαριστούμε, Ιζαμπέλα Ντεμόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα όλα να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Ίστραν για το σχέδιο της έκθεσης. Νομίζω ότι είναι πλήρες το κείμενο και εγώ, με πιο συγκεκριμένα νομίζω ότι έχει τη σωστή κατεύθυνση γιατί πρόκειται για ε, μια κατεύθυνση που θα πρέπει να την ακολουθήσουμε χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι. Μιλούμε για την Ευρώπη ως προορισμό. Και πρόκειται για πάρα πολλούς υπεύθυντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πρόκειται για έναν τουρισμό που είναι μια μεγάλη αγορά. Μεγάλη αγορά είναι και οι τρίτες χώρες. Ε, και ε, αυτή η κυκλοφορία προς εμάς θα αυξηθεί Οπότε δεν θα πρέπει αυτό να το παραλείψουμε γιατί είμαστε ο πρώτος ε, παγκόσμια προορισμός και αυξάνεται μέσα στον χρόνο περνά ο τουρισμός. Έχουμε βέβαια και άλλους προορισμούς που είναι ανταγωνιστές μας γιατί και για αυτούς αυξάνεται ο τουρισμός. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, πώς θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία και Αντίστοιχα θα πρέπει να είναι και η νομοπαρασκευαστική διαδικασία, μείωση του κόστους, απλούστευση. Επίσης, θα πρέπει να δείξουμε και κάποια αλληλεγγύη ε, προς τα υπόλοιπα κρατή μέλη. θα πρέπει να ε, διευκολύνουμε τόσο πάντων την πρόσβαση. Είναι βέβαια σημαντική και η ασφάλεια έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές έρχονται έτσι ε, τρομοκράτες. Σωστά τα είπατε για την ε, Κίνα. Επομένως έχουμε αυτές τις ε, πτήσεις, όμως θα πρέπει η Ένωση να έχει ένα μάρκετινγκ πιο αποδοτικό, γιατί είναι παγκοσμίως προορισμός. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το, παραδείγματα παραδείγμα των που έχουμε, που έχουν κάνει άλλοι. Έχουμε πίεση χρόνου, παρακαλώ την Κομισιόν να συντομεύει και στο τέλος ο εισηγητής. Η κυρία Γιολάντα Καζέγο Γκαλίντα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή αλλά και τους υπόλοιπους βουλευτές επειδή βοήθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την πρόταση, με αυτή τη δέσμη μέτρων. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε τώρα να θεωρηθεί αυτό το καθεστώ και η πολιτική μα για τι θεωρήσει, ώστε να μπορέσουμε να απλουστεύσουμε τι διαδικασίε, να γίνουν όλα ταχύτερα, να φέρουμε έναν, ε, μια εναρμόνιση και έτσι να ελκύσουμε περισσότερου νόμιμου ταξιδιώτε, αλλά και να αλαφρύνουμε και το βάρο των προξενείων. ο τουρισμό βοηθάει στην δομική ανάπτυξη και οι ρυθμίσει πάλι των θεωρήσεων. Ε, ταυτόχρονα προσπαθούμε να καλύψουμε ένα βασικό στόχο τη πολιτικής θεωρήσεων. Να σταματήσουμε τη λαθρομετανάστευση και να έχουμε ασφάλεια στην περιοχή Σέγγεν. Άρα πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ αυτών των δύο στόχων. Ασφάλεια αλλά και προσπάθεια διευκόλυνσης νομίμων ταξιδιών προ την Ευρώπη, αλλά βοηθήσουμε την για ανάπτυξη. Τώρα, όσον αφορά αυτή την, ε, τη θεώρηση περιφορά, ε, είπαμε ότι έχουμε αυτούς τους ξένους που θα μείνουν 90 χρόνια, 90 μέρες συγγνώμη, ε, όχι στους αμυγιστικά σε ένα κράτος μέλος, να έχουμε εναρμονισμένη προσέγγιση. και επίση αν θα γίνουν τι διμερεί σύμφωνε που έχουν κάποια κράτη-μέλη με τρίτε χώρε. Ε, και εκεί σε αυτέ τι περιπτώσει δεν χρειάζεται βίζα. Οπότε έχουμε διαφορετικού κανόνε για διαφορετικού ε, επισκέπτε ανάλογα με τι ρυθμίσει με τι χώρε του αντιστοίχω. Επομένω, η πρότασή μα ισορροπεί μεταξύ όλων αυτών. Ευχαριστούμε για τι παρατηρήσει, ιδίω του εισηγητή Ευχαριστούμε τις τροπολογίε και πολύ σωστό αυτό το να υπάρχει ένας άλλος φορέας να χειρίζεται τις θεωρήσεις και όχι αναγκαστικά αυτό να περνάει από το προξενείο. Επίσης, όσον αφορά τον προβληματισμό για την ασφάλεια. Για αυτές τις ε, ε με αυτές τις θεωρήσεις τέλο πάντων περιφόρα, οπότε είπαμε ότι θέλουμε την ασφάλεια στην περιοχή Σέγγεν και υπάρχουν προϋποθέσεις όσον αφορά αυτές τις καινούργιε θεωρήσει. Είναι πιο αυστηροί οι κανόνες ε, από ότι παλαιότεροι ενία οι Και κάποιο για να παρακάμψει το σύστημα θα έπρεπε να κάνει κλασική αίτηση ε, γιατί σα είπα, οι κανόνε για τι καινούργιε είναι πιο αυστηρέ. Τώρα, όσον αφορά την προσέγγιση για την ε, διευκόλυνση, όσον αφορά αυτό το μητρό των ε, συχνών επισκεπτών και ταξιδιωτών, είπαμε ότι έχουμε πολλέ βίζε ε, εισόδου και την προηγούμενη εφαρμογή του πλαισίου ε, του νομοθετικού είναι καταγεγραμμένες αυτές οι βίζες εισόδου, έτσι κι αλλιώς. Επίσης ε, αναφέρθηκαν και οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Εμείς ήδη έχουμε τοποθετηθεί στην Επιτροπή σα και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και θεωρούμε ότι αυτές οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις θα πρέπει να ρυθμιστούν εκτός ενωσιακού κώδικα. Πρόκειται για κάποιους που δεν έρχονται για σύντομο διάστημα. Έρχονται για να μείνουν περισσότερο. Χρειάζονται διεθνή προστασία. Άρα είναι θέμα το επαναγκατάσταση με την κατάσταση κλπ. Το θέμα τώρα της εκπροσώπηση. Έχουμε και εδώ κάποιες ε, τροπολογίες του εισηγητή. Στην πρότασή μας λέμε να είναι υποχρεωτική εκπροσώπηση. Δηλαδή, να μπορούν όλοι να βγάλουν την αίτηση στην χώρα διαμονής, να μην χρειάζεται να ταξιδέψουν. Όμως, δεν ισχύει αυτό σήμερα. Έτσι λοιπόν θα είναι ευκολότερη η υποβολή της αίτησης. Επίσης έχουμε και αυτούς που θα παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, τους νέους αυτούς φορείς και θα είναι πιο εύκολο στον κόσμο να υποβάλει αίτηση. Επίσης, είπαμε θα πρέπει να παρακολουθούμε το έργο αυτών των παρόχων αυτών των υπηρεσιών. Τώρα για το χρόνο βολής αίτησης μιλάμε για τρεις μέχρι έξι μήνες. Μέχρι δώδεκα, είπε ο εισηγητής. Ίσως αυτό είναι πολύ, γιατί παρά είναι μακρό διάστημα για να μπορέσει κανείς να παρακολουθήσει την κατάσταση του ετούντος γιατί μπορεί να έχει αλλάξει η οικονομική του κατάσταση σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε για τι τροπολογίε και ευχαριστούμε για τη στήριξή σα στην πρότασή μας. Ευχαριστώ και πάλι ο εισηγητή ο Ιστβάν Χέιλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφου μου για την υποστήριξή τους και τις προτάσεις τους. Πορτογαλία, Ισπανία, Φιλανδία, Ιταλία. Χώρες που ανήκουν στην ζώνη του Σέγγεν από διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Όλοι υποστηρίζουν την πρόταση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω την Κλαβδία παραδείγματος χάρη, την Ντουμπράβκα και για την δική σας υποστήριξη από την Κροατία, τη Ρουμανία, από χώρες εκτός Σέγγεν και εγώ βέβαια είμαι Ούγκρος και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευρύνουμε τα σύνορα του Σέγγεν και να είμαστε ενωμένοι προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά που είπατε, για την ιστοσελίδα. Χαίρομαι που θέσατε το θέμα αυτό, το όρο θέμα των αιτήσεων από το ίντερνετ, το είπαν πολλοί συνάδελφοι και θα προσπαθήσω να το τονίσω περισσότερο στους επόμενους μήνες. Συμφωνώ και με τον κύριο Ντάλτον, δεν το ανέφερα σε εκτενές επίπεδο πρέπει να έχουμε σαφήνεια, ασφάλεια, ένα ασφαλές σύστημα, σύμφωνα μαζί σας. Αυτή είναι η βασική αρχή, βέβαια. Αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως πρόσχημα την ασφάλεια για να μην κάνουμε μεταρρύθμιση αυτών των κανόνων. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, οποιοδήποτε από εσά μπορεί να τροποποιήσει, να βελτιώσει τις προτάσεις αυτέ να κάνετε περαιτέρω προτάσεις μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω ότι θα έχουμε περαιτέρω προτάσεις. Θα είμαι σε διακοπές, αλλά στην Ουγγαρία θα είμαι σε επαφή μαζί σας. Μπορείτε να μου στείλετε email και πείτε και στου συναδέλφου σας Και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο θα τα προετοιμάσουμε αυτά. Νομίζω ότι και οι εκπρόσωποι άλλων φορέων από άλλες επιτροπές θα μπορούσαν να είναι εδώ. Ε, εντάξει, καλοκαίρι είναι, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ λοιπόν. 8 Σεπτεμβρίου είναι προθεσμία για τις τροπολογίες. 10 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε και μετά θα ακολουθήσει η Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ και ερχόμαστε στο λουκούμιο σημείο της ημερησίας διάταξης, την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για την εσωτερική ναυσιπλοεία στην Ευρώπη και η, η Ιβάνοβα είναι η αρμόδια από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Την ευχαριστώ που είτε και της δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ, μιλάτε και γερμανικά. Αξιότιμοι βουλευτέ, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση και πάντοτε χαίρομαι όταν έρχομαι στην Επιτροπή σα. Πριν από λίγου μήνε παρουσίαση την ειδική έκθεση για την ε, για αστικές μεταφορές από πλευρά του Ελληνικού Συνεδρίου και σήμερα χαίρομαι που μου έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για τις εσωτερικές ε, ε πλωτούς οδούς. Ε, δυστυχώς από το 2001 και μετά, όπως λέει και ο τίτλος έκθεση, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές. Ε, ξέρετε ότι είναι, πρόκειται για ένα από τους τρεις βασικούς τρόπους ε, μεταφορών, 30.000 περίπου χιλιόμετρα εσωτερικών πλωτών οδών ε, σε ένα ποτάμι μπορούμε εκατοντάδες φορτηγά να να αντικαταστήσουμε με ένα μόνο πλοίο, ε, μειώνοντας τις εκπομπές, ε, τα ατυχήματα, τη συμφόρηση τη, και από το 2001 και μετά άρχισε να προωθεί ε, τι δασταρική πρωτοσυλλογέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτού ακριβώς ακριβώ λόγους λόγου και έχει εντοπίσει τα σημεία συμφόρηση που είναι και τα βασικά εμπόδια για αυτόν τον τρόπο μεταφορών. Για την περίοδο προγραμματισμού το 2013 ε, έχουμε χρηματοδότηση από τα ΔΕΛΕ 747 εκατομμυρίων και 531 εκατομμύρια από τα διαστατικά ταμεία για μελέτες και για προγράμματα βελτίωση των υποδομών. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες αναμυσιπλοείας, ε, αυξάνοντας το ύψος ε, ε, των γεφυρών, παραδείγματος χάρη, βελτιώντας τη συνεργασία των εθνικών αρχών, ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τα συνοριακά τμήματα και εμείς αποτιμήσαμε σε αυτόν τον τομέα των στρατηγικών αν υπάρχει ικανοποιητική και γι' αυτό επιλέξαμε 12 προγράμματα για επιτόπια επιθεώρηση σε 4 κράτη-μέλη, Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία και Ζαρία. 88% των ε, δαπανών ε, των προγραμμάτων ε, για την περίοδο 2007 έως 2013 ήταν σε αυτές τις τέσσερις χώρες. Σε αυτό το έλεγχο επίσης αναθεωρήσαμε την πολιτική που εφαρμόστηκε από το 2001 και μετά. Είχαμε συνεντεύξει με συμπλεκόμενου φορεί από τιμή των προγραμμάτων και επισκόπηση των βασικών δικτών ε, σε σχέση με τα μοντέλα για την κοινή ναυσιπλοεία. για τη μετατόπιση ε, των μεταφορών από τις οδικές μεταφορές στις εσωτερικές πλωτούς ε, οδούς και τη βελτίωση της επιλογιμότητας. Βλέπουμε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Ε, το μοντέλο επιμερισμού βλέπουμε από το 6,4 έχουμε βελτιώσει τα ποσοστά ανεβαίνοντα το 6,7% αλλά δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι αυτό συνδέεται με παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο 6 βασικά σημεία συμφόρηση έχουν αρθεί και ε, κατά πόσα πιθανότητα θα χρειαστούν 60-70 χρόνια για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα σημεία συμφέρουσης που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης ε, ε, η μεταφορά εμπορευμάτων έχει επηρεαστεί σε πολύ μικρή κλίμακα διότι άλλα παρακείμενα σημεία συμφόρησης δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Επίσης εξετάσαμε τα προγράμματα βελτίωση των υποδομών όμως ε, βλέπουμε ότι ε, δέκα μόνο ε, είχαν μια θετική συμβολή, ενώ άλλα έξι ήταν εν τέλει. Και στο εγγύς μέλλον δεν πρόκειται να έρθουν τα σημεία συμφέρουσης. Ε, Χρησιμοποίησαμε ως υπόδειγμα τρία προγράμματα για να δούμε αν έχει βελτιωθεί η πλοημότητα. Δύο προγράμματα σχετίζονταν με τον τουρισμό και είδαμε ότι ούτε καν ασχολήθηκαν σε αυτά τα προγράμματα με τα σημεία συμφόρηση. Αναλύσαμε και τις στρατηγικές άλλο με το ελέγχο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδαμε ότι οι στρατηγικές ε, δεν βασιζόντουσαν σε ε, ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία και ανάλυση δεδομένων, οπότε ε, το αποτέλεσμα ω προ την βελτίωση των υποδομών και τη μετατόπιση των μεταφορών προ τι εσωτερικέ πλουτοσυδρού είναι κάτι που ουσιαστικά μα είναι άγνωστο. Ε, στη συνέχεια, ο επιμερισμό των μεταφορών στου διάφορου διαδρόμου είναι κάτι που επίση μα είναι άγνωστο, διότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για το μοντέλο επιμερισμού της ε, ε, βελτίωσης ε, της ε, πλοημότητας. Επίσης, δεν αντιμετωπίσαμε τα βασικά εμπόδια. Υπάρχουν ανακολουθήσει ανάμεσα στις εθνικέ στρατηγικές. Χάσμα χρηματοδότησης ανάμεσα στο εκτιμόμενο κόστος για την άρση όλων των εντοψέτων σημείων συμφόρησης και των διαθέσιμων πόρων χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, η προστασία του περιβάλλοντος ε, δεν συνάδει με τη μετατόπιση των μεταφορών προς εσωτερικές ε, πλωτές οδούς και δεν υπάρχει παρκή συντήρηση των ποταμιών, των υποδομών στα ποτάμια. Κάναμε δύο βασικές συστάσεις για δύο διαφορετικές επιτυχίες που καλύψαμε στην έκθεσή μας, οι επιδόσεις, τα αποτελέσματα των προγραμμάτων ως προς τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εσωτερικές πλωτές οδούς για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της ε, χρηματοδότησης. Για αυτό το είδο μεταφορών προτείνουμε ε, να ε, αποδοθεί προτεραιότητα από πλευρά των κρατών μελών στα προγράμματα που έχουν τα πιο άμεσα θετικά αποτελέσματα και να έχουν και ένα πιο αποτελεσματικό πρώτερο σχεδιασμό για την καταπολέμηση των σημείων συμφόρηση. Για το συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λύσει τα θετικά αποτελέσματα των μεταφορών σε ιστορικέ πρωτεύουσε στα διάφορα τμήματα του ποταμού και να τα συνδυάσουμε με τι εκτιμήσει που έχουν γίνει με τα ΔΕΔΕ και συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν κάποιοι μη υλοποιήσιμοι στόχοι από πλευρά των κρατών μελών για την καταπολέμηση των σημείων συμφόρηση και θέλουμε να ενισχύσουμε επίση την νομική βάση ώστε να διευρύνουμε ε, τι ε, υποχρεώσει ε, υποβολή αναφορών σε σχέση με την πλοημότητα των διαφόρων τμήματων ποταμών και να βελτιωθούν και τα προγράμματα με πιο συντονισμένο τρόπο για την συντήρηση των υποδομών των ποταμών. Ε, με αυτέ τι τράσει ελπίζουμε ότι θα έχουμε πιο αποτελεσματικέ και πιο ποιοτικέ ε, μεταφορέ στι ιστορικέ πρωτεύουσε. Πριν από λίγε εβδομάδε ε, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Επιτροπή για αυτό το θέμα. κύριε Νοβακόφ, σα λέγω είστε εισηγητής. Θέλω να σα συγχαρώ. Πολύ εξαιρετικό, εξαιρετική ποιότητα το πρόγραμμα το σχέδιο εργασία που έχετε καταρτήσει. Ελπίζω να σα βοηθήσουμε στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και ω συνήθω ε, είμαστε στη διάθεσή σα ε, για επικοδομητικέ και καρποφόρε συζητήσει. Εμεί σα ευχαριστούμε για την παρουσίαση και ε, θεωρώ πολύ καλό ότι γίνονται τέτοιε αναλύσει και κυρίω ότι μπορούμε να τη συζητήσουμε σήμερα. Δυστυχώ δεν είναι αθρώα η προσέλευση, αλλά αυτοί που είναι εδώ ενδιαφέρονται και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την παρουσίαση και κύριο κύριος στο θα πάρει το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ευχαριστήσω τον ε, την πρώην μας ε, που ήταν μα στο ΕΛΠ, η κυρία Ιβανόβα, ήρθε να μα ξαναδεί σήμερα. Και πρέπει όμω να τονίσουμε το ότι κάθε από εδώ με στεναχωρεί. Την τελευταία φορά που μα επισκέφτηκε, η κυρία Ιβανόβα ήρθε με μια πολύ αυστηρή έκθεση. Πολύ επικριτική λοιπόν και αφορούσε την κινητικότητα της πόλης. Και σήμερα λοιπόν ήρθε και μας καθίζει πάλι στο σκαμνί. Επικρίνει αυτά τα οποία έχουμε κάνει με τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Βέβαια δεν έχει και πολύ άδικο. Μα αυτή είναι η δουλειά της. Αυτή είναι η δουλειά του Ελληνικού Συνεδρίου. Να εξετάζει το τι συμβαίνει και να επισημαίνει τα στραβά. Είπατε στην εισήγησή σα ότι αν ε, πρέπει να δαπανίσουμε ε, νέους πόρους, αυτό χαροποιεί πάντοτε όλο τον κόσμο, όμως μετά υπάρχει το άλλο θέμα της υπευθυνότητας. Είναι τώρα δύσκολη ώρα που έχει περάσει η ημέρα, αλλά χρειαζόμαστε φρέσκο χρήμα. Και πρέπει να δούμε βέβαια πώς ε, αξιοποιούνται αυτά τα κονδύλια και ξέρετε στα Ολλανδικά ΜΜΕ ήλκησε όταν πρωτοβγήκε αυτή η είδηση μεγάλο ενδιαφέρον. Είδαμε ότι αυτό γίνεται και σε πολλά κρατημέλη έχουμε ένα σωρό ε, μικροπρογράμματα, μικροσχέδια, μικροέργα, έχουμε αυτούς τους υδατοφράκτες, έχουμε και πάρα πολλά στοιχεία ε, διασυνοριακότητας, αυτά που μας αναφέρονται. Και δεν ξέρω μήπως κάτι παρεξήγησα όπως είπατε, αλλά νομίζω ότι είπε η κυρία Ιβανόβα ότι όλα αυτά σχετίζονται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Εγώ όμως θεώρησα ότι ο έλεγχος που έγινε από το συνέδριο έγινε κατόπιν. Αφού δηλαδή είχε, έχει τελειώσει η υπόθεση των διευρωπαϊκών δικτύων. Αν όλα αυτά περιέχονται, υπάγονται τέλο πάντων στο καθεστώ των διευρωπαϊκών δικαιών, καλώ, καλά τα πήγε το Ελληνικό Συνέδριο. Όμω, εμεί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θεωρούμε ότι αυτή η υπόθεση ανάγεται στην περίοδο πριν εγκριθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και αυτό αφορά τι προτεραιότητέ μα για αυτού του διαδρόμου και σε σχέση με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της ε, λευκη βιβλου Βίβλου είπαμε ότι πήγαμε 6,4-6,8 ε, τα οποία είναι φραγκοδίφραγκα, άρα δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Τι να σα πω κύριε Ιβανόβα. Είναι μεγάλη η δυσαναλογία Επομένως ελπίζω ότι όλα αυτά που τώρα εξετάζουμε αφορούν τη χρονική περίοδο πριν τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Άλλο θέμα. Συνεχίζει το Ελληνικό Συνέδριο να παρακολουθεί, να ελέγχει τι γίνεται τώρα. Ωραία, έχουμε εδώ την εκθεσή σας, θα την ε, μελετήσουμε για να μάθουμε. Αλλά και του χρόνου τα ίδια θα γίνουν. Δεν θέλουμε να πάρουμε ένα τέτοιο κατήφορο. Εγώ αποδέχομαι τα συμπεράσματά σα. Να δούμε τι θα πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν ξέρω πω δεν φταίμε εμεί. Άρα, ξεκαθαρίστε σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεστε, πριν ή μετά τα δέδα. Και μετά να δούμε τι έγινε με τη δαπάνες από τότε που ε, συνετάγει αυτή η έκθεση. Οπότε για να δούμε τώρα πώς να τον βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ, η Μάγια Κίλενεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε, σας ευχαριστώ για την ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ την κυρία Ιβάνοβα για την έκταση αυτή που απαιτεί από εμά το Κοινοβούλιο να κοιτάξουμε στον καθρέφτη και να σκεφτούμε αυτά τα οποία πήραμε υπό μορφή ανάδρασης από το Ταμείο από το Ελεκτικό Συνέδριο και από τους φορείς μεταφορών για το αν τα χρήματά μας πιάσανε τόπο και αν έχουν χρησιμοποιηθεί λογικά. Έχουμε κοινούς στόχους. Είναι οι στόχοι μας να δημιουργήσουμε ένα κοινό σύστημα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα είναι απλώς ένας εμβαλωματικός καμβάς και τελικά δεν θα έχουμε πετύχει το στόχο μας. Και επειδή ο κύριος Φαντεκάμπ είναι πάρα πολύ στεναρός υπέρμαχος των ε, εσωτερικών ιδιαίτερων δρόμων, θα ήθελα να τον υποστηρίξω από τα αριστερά. Να βρούμε στόχους, λογικούς στόχους, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το χρήμα του φορολογούμενου με ένα θετικό τρόπο για να βελτιώσουμε την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουμε για τις μεταφορικές μας ανάγκες στο μέλλον που περιλαμβάνει τους εσωτερικούς υδάτινους του Κόβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για το έγγραφό της, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είχα την ευκαιρία του το επεξεργαστώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι δεν είναι μια εκθέση του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι μια σημαία που ανεμίζει και αναπετάνεται μπροστά στα μάτια μας. Γιατί δείχνει την κατάσταση στις εσωτερικές υδάτινες οδού. Είναι ένα σημαντικό τομέα για την ευρωπαϊκή πολιτική και στα θέματα συνοχής. Έχουν ταπανηθεί δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές, σημαντικά σημεία συμφόρησης. Πολλές φορές λόγω έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας των, των ε, εθνικών υπηρεσιών χρειαζόμαστε περισσότερα σχέδια. που έχουμε χρειαζόμαστε περισσότερα σχέδια σύνδεσης με τους κύριους διαδρόμους, με τα σχέδια που έχουν ήδη εγκριθεί στα κάτι μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού εμείς δώσαμε έμφαση σε θέματα όπως πραγματικά η βελτίωση του, της πλοημότητας του Δούναβη, γιατί αυτός είναι κύρια εσωτερική οδός. Έχουμε περιοχές που είναι πιο βαθύς και πιο φαρδής ο Δούναβης, ώστε να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα πλοία, χρειάζεται να έχουμε πιο ψηλές γέφυρες για να περνούν τα φορτηγά ενώ στο επόμενο κράτος δεν γίνεται τίποτα. Το πλοίο πάει μέχρι ένα σημείο και μετά κολλάει. Είναι σαν να έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει μόνο ένα αεροδρόμιο. Πετάει το αεροπλάνο και δεν μπορεί να προσγειωθεί πουθενά, πρέπει να γυρίσει πίσω. Στράφει πάει το αεροδρόμιο, στράφει και το αεροπλάνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερο συντονισμό και θα χρειαστεί να ενισχύσουμε και το ρόλο της Κομισιόν όταν εγκρίνονται αυτά τα σχέδια και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τα κράτη-μέλη να έχουν καλύτερο συντονισμό από ότι τώρα και μετά η χρήση των κονδυλίων από το Connecting Europe Facility και τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι απαραίτητη. Αυτή η έκθεση λοιπόν θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε όχι μόνο αυτό το τομέα της πολιτικής συνοχής, αλλά όλους τους τομείς της πολιτικής αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ως τελευταίος εγώ ο ίδιος. Εμένα δεν με εκπλήσει αυτό που λέει η έκθεση, είναι πολύ σημαντική. Η δική μου εμπειρία είναι ότι στα θέματα των εσωτερικών ε, υδατήρων οδών υπάρχει ένα τεράστιο όνειρο το και όραμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα 80% της ε, εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη είναι στον Ρήνο. Αλλά 90% των χρημάτων πηγαίνουν για να υποστηρίξουν διάφορα οράματα. Αυτό δεν έχει νόημα. Στη Γερμανία ο αριθμός των πλοίων έχει μειωθεί και ο ρόλος της εσωτερικής ναυσιπλοείας έχει κατέβει το 20% στα 8%. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Γιατί γίνεται αυτό. Η δική μου πεποίθηση είναι ότι δεν έχουμε αρκετά πυκνό δίκτυο σε σχέση με τις συνδρομικές ιωδικές συνδέσεις και φυσικά λόγω της ε, μορφολογίας του εδάφους δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει παντού η εσωτερική ναυσιπλοεία. Και εκεί που είναι δυνατόν δεν χρησιμοποιείται. Δεν έχει λοιπόν νόημα να λέμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε τον Έλβα και το Δούναβι κτλ. Από το Ingolstadt στην Μαύρη Θάλασσα λέγανε πριν από χρόνια ότι θα μπορέσει να κινείται ένα πλοίο. Όταν έρχεται όμως το ένα μεγάλο πλοίο ε, και αντιμετωπίζει ένα άλλο πλοίο είναι πολύ δύσκολο να περάσουν και τα δύο. Εγώ πήγα 100 χιλιόμετρα με ποδήλατο στο Δούναβι είδα τουλάχιστον τρία πλοία. Αλλά πολύ λίγα είναι τα πλοία τα οποία μπορούν να περάσουν από τα πλοία τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Έχουν πρόβλημα με το βάθος. Τα πλοία τα οποία μπορούν να πάνε στον Δούναβη παρόλα αυτά δεν πηγαίνουν και αυτά. Εξακολουθούν τα οράματα αυτά για τον Δούναβη και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είπε δεν θα κάνουμε διεύρυνση του Δούναβη στη Βαβαρία, ενώ οι θέλουν να υπάρξει ανάπτυξη. Οτιδήποτε λοιπόν γίνεται προσπάθεια να γίνει μετά από 30-35 χρόνια δεν προχωράει και η δική μου πεποίθηση ως Γερμανού είναι η εξή. Για κάθε πλοίο που πλέει σε εσωτερικές υδάτινες οδούς χρειαζόμαστε τρεις γραφειοκράτες. Κάθε νέο σχέδιο δεν δημιουργεί τίποτα οι πολιτικοί ερχόνται και λένε θα πρέπει να φέρουμε τους ε, διοικητικούς για να αναλάβουν τις αρμοδιότητές τους. Αλλά με τον τρόπο αυτό δεν καταφέρουμε να προχωρούμε. Τρεις διοικητικοί πάλι αναπλοίο. Αναμαούνα δηλαδή. Δεν υπάρχει, έχουν μεγάλα πλέον δεν πληρώνουν φόρο στα καύσιμα όπως και άλλες μορφές μεταφορών. Αλλά δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά με τις άλλες μορφές. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν μπορεί κανείς με επιδοτήσει μόνο να το πετύχει στο Βερολίνο. Όταν έπεσε το τείχος θέλαμε να πάμε στον Όντερ και αλλάξαμε τους υδατοφράκτες στο Βερολίνο. Ο αρμόδιος Υπουργό μεταφορών στο κρατήριο του Βερολίνου είπε βεβαίω έχουμε φτιάξει τους υδατοφράκτες ώστε να περνούν να μπαίνουν μεγάλα πλοία. Αυτό είναι επένδυση για το μέλλον, δεν έχει να κάνει με το τώρα. Και το είπε ο εκπρόσωπο για τον, ε, της λε είπε είναι σημαντική η υδατοφράχτες γιατί οι σιδηρόδρομοι από το Βερολίνο στην Βαρσοβία είναι μόνο εν μέρη έτοιμη η γραμμή. Και είπε επομένως έχουμε μια προοπτική και εγώ γέλασα γιατί πραγματικά αυτό δεν έγινε πραγματικότητα και επειδή βλέπω τον κύριο Φέρμπερ αναφέρομαι στο, στη σύνδεση Ρήνου Δούναβη. Αυτό το κανάλι υποτίθεται ότι θα ε, είχε μεγάλη κίνηση, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα και το 10% αυτού που προβλεπόταν ερχόταν. Ήταν ένα σχέδιο λοιπόν το οποίο κόστισε δισεκατομμύρια και είπε ότι ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών της Γερμανίας ήταν από τις μεγαλύτερες βλακίες που έχουν ποτέ γίνει. Θα μπορούσε κανείς να το φτιάξει λοιπόν πολύ πιο φθηνά αυτό. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Δεν θέλω λοιπόν να διαφυσβητήσω αν υπάρχουν κενά ή σημεία συμφώσεις. Αλλά το να έχουμε συνέχεια οράματα όταν βλέπουμε νερό ότι θα έχουμε μεγάλα πλοία. Ποτέ δεν θα πετύχει αυτό. Είναι λάθος και πρέπει να πούμε stop κάποια στιγμή γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για πιο σημαντικά σχέδια. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με λίγα λεφτά και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή να λάβουμε το λόγο από την πλευρά της του Ελεκτικού Συνεδρίου. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και για αυτή σας την εισήγηση. Όμως, να, με όσα είπατε, σας εγγυώμαι ότι πρόκειται το ελεγκτικό συνέδριο να σας απευθύνει καινούρια έκθεση. Γιατί εξηγήσατε τόσα πολλά. Είπατε τόσα πολλά για το, το, το, θέμα μας, την προβληματική μας για το εσωτερικές πρωτές οδούς που τι να πω. Καλά εντάξει τώρα πέραν των αστείων. Ε, είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον Συνέδριο η έκθεση. Θέλουμε ότι είναι αξιόλογη, δεν μα έρθει ο τίτλο, αλλά δυστυχώ τη σήμερα ημέρα πρέπει κανεί να, να είναι ευρηματικό με τον τίτλο για να μπορέσουν να τον δημοσιεύσουν εφημερίδε και ΜΜΕ. Γιατί δεν θεωρούμε ότι υπάρχει αντιστοιχία με το περιεχόμενο τη έκθεση. Οπότε και νομίζω πω συμπερασματικά είναι μια καλή έκθεση. Νομίζω ότι προβλέψαμε πολλές εξελίξεις τότε. Όχι, δεν μιλάμε μόνο για προγράμματα ε, ΔΕΔ. Είναι πολύ λίγα από αυτά το δικτυό Συνέδριο, πάρα, πολύ θετικά βλέπει αυτά που καλύπτονται από τα διευρωπαϊκά Όμως τώρα, τώρα έχουμε καινούργιο τοπίο καινούριο καθεστώς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουμε και τα περιφερειακά ταμεία και άρα έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν, να προτείνουν τα κρατημέλη. Όχι, όχι, δεν υπήρχε κάποια στρατηγική σε σχέση με την στάση μας. Θα προβάλλουμε του παρελθόν, οπότε με του συναδέλφου, και Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική, προσπαθούμε πάρα πολύ σοβαρά να δούμε τι θα κάνουμε με τα καινούργια μέσα πολιτικές και να μπορούμε να βγάλουμε ζουμί από ό,τι έχουμε στη διάθεσή Άρα, το θέμα δεν είναι ότι θα υπήρχε διασπάθηση των πόρων, αλλά είναι τόσο μεγάλη η οικονομική στενότητα, ούτω ώστε ότι θα έπρεπε να γίνει καινούργια εκταμίευση για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλο αυτό το δίκτυο των εσωτερικών Κύριε Φαντεκάμπ, σας ε, υπόσχομαι ότι θα ακολουθήσει νέα έκθεση πέραν των αστείων σε σχέση με όλα αυτά που αναφέρει η έκθεση και θα συνεργαστούμε με τους συναδέλφους και στο Ελληνικό Συνέδριο και με τους ε, συνάδελφους ευρωβουλευτές. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η Λιάννα Ιβάνοβα έχει τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου για όλα τα χρήσιμα και πολύτιμα σχόλια τους. Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Μας βοηθούν και μας να βελτιώσουμε την ε, εκθεσή μας. Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάμ για τις εκθέσεις. Είπα την τελευταία φορά ίσως ήμουν πολύ ευγενική προς τη Δομησιόν. Αλλά κατανοώ αυτό που είπατε ότι ίσως είναι κάπως αρνητικός ο τίτλος της έκθεσης. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όχι να είμαστε αρνητικοί για να είμαστε αρνητικοί, να είμαστε επικοδομητικοί αντίθετα, να δείξουμε πού είναι οι δυσκολίες και τα σημεία που υπάρχουν ελλείψεις και να βελτιώσουμε τα πράγματα. Για να έρθω τώρα στα ερωτήματά σας, δεν είναι μονάχα τα σχέδια τα διευρωπαϊκά που είδαμε, Είδαμε και σχέδια περιφερειακού ταμείου, ιδίως στο διάστημα 2007-2013, είναι μακροχρόνια σχέδια και για κάποια από αυτά περιμένουμε ακόμα να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτή είναι η χρονική περίοδος η οποία καλύφθη και μπορεί στη συνέχεια μετά και από αυτή τη συζήτηση, όπως πήγε μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συνέχει, μια έκθεση συνέχειας. Ξέρουμε το 2010 οι κατευθυντές γραμμές των ε, διευρωπαϊκών του 2010 ήταν μια απόφαση η οποία δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη. Οι νέες τώρα αποφάσεις έχουν τη μορφή κανονισμού, επομένως απορρέουν άμεσα αποτελέσματα για τα κράτη-μέλη και με τους νέους αυτούς κανονισμούς υπάρχει ένα, ένας πυρήνας και ένα συνεκτικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η Κομισιόν και διαδρόμους για τους οποίους υπάρχουν συντονιστές και προβλέπεται και μια πελετέρω μελέτη για το 2015 για να υπάρξει μέσα στο 2015 να έχουμε μια πιο βαθύτερη ανάλυση. Εμείς όμως ως ελεγκτές κοιτάμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το σύνολο των αποτελεσμάτων, όπως σας είπα θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να δώσουμε συνέχεια. Κυρία Κίλλονεν αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για την θέσπιση κοινών στόχων και τα μεμονωμένα κομμάτια του παζλ. Εκεί βλέπουμε να υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, έχουμε προβλήματα διάσπαρτα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει πάντα κάποια επικοινωνία και κάποιο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να μπορέσουν τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπιστούν με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Και για σας κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην έλλειψη πυκνών δικτύων στις, ε, στους εσωτερικούς υδάτινους δρόμους και γι' αυτό το λόγο μία από τις ε, συστάσεις μας είναι τα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε σχέδια εσωτερικών υδατινών δρόμων που έχουν δυνατότητα άμεσου ωφέλους. Μόνο αυτά τα οποία έχει πραγματικά νόημα να υποστήριξει κανείς με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο για να ευνοήσουμε την δημοσιογραφική μεταφορά. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και προσβλέπω την περαιτέρω συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μία παρατήρηση και μόνο. Η Κομισιόν επέκρινε τον τίτλο, όχι το περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο η Επιτροπή μας τον τίτλο επέκρινε. Συμφωνούμε όμως απόλυτα στο περιεχόμενο. Είμαι πραγματιστής. Άμα το περιεχόμενο είναι σωστό και όχι ο τίτλος δεν πειράζει. Το αντίθετο θα ήταν πρόβλημα. Επίσης, μια δεύτερη παρατήρηση, πρέπει να μάθουμε από τα σφάλματά μας. Γι' αυτό είναι καλή η έκθεση, γιατί αναφέρει τις περιπτώσεις όπου αστοχήσαμε και ένας καλός μαθητής, ο πιο καλός ο μαθητής δεν κάνει δύο φορές το ίδιο λάθος. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει να πάμε. Και επειδή είναι και η τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις διακοπές, σας εύχομαι όλους καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, γυρίστε υγιείς και με καλή διάθεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας μετά τις διακοπές. 31 Αυγούστου. 5 η ώρα. 5 η ώρα. Είμαστε η πρώτη επιτροπή που, συνεχίζει μετά τις διακοπές. Που αρχίζει μετά τις διακοπές. Ευχαριστώ. Καλές διακοπές.